Ladies and gentlemen, please be seated. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε την απογευματινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας. Τρία πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα θα καλύψουμε σήμερα το απόγευμα. Ξεκινήσουμε λοιπόν χωρίς καθυστέρηση. Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να σας παρουσιάσω το επόμενο σημείο που έχουμε στη μερίσια διάταξη, προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας, στρατιωτικοποίηση της περιφέρειας του Καλίνιγκραντ. Καλίνιγκραντ Όμπλαστ, επαρχία του Καλίνιγκραντ, όπως το αποκαλούν. Έχουμε τρεις πολύ διακεκριμένους ομιλητές μαζί μας σήμερα. Θα ήθελα καταρχάς να σας παρουσιάσω τον συμπατριώτη μου, τον κύριο Ιώτρε Παχόλσκι, ο οποίος είναι αναπληρωτής διευθυντής στο Υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας και είναι υπεύθυνο για ζητήματα διεθνούς άμυνας και ασφάλειας. Στα αριστερά μου κάθεται ο Διευθυντής ε, του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Επιχειρήσεων της, ε, του Υπουργείου Άμυνας της Λιθουανίας, ο κύριος Ντέιβις ε, Πετραίτης, και στη συνέχεια, πιο πέρα στα αριστερά μου πάλι, έχουμε τον επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής Άμυνας και Σχεδιασμού, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, τον κύριο Γκάμπριελ Μπερνιέ. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αποστολής μας στην Ουκρανία και κατά τη διάρκεια των επαφών που είχαμε με σημαντικούς παράγοντες ε, εκεί, σε όλους τους κλάδους της κυβέρνησης, αλλά και σε επαφές που είχαμε με διοικητές, στρατιωτικούς και με μέλη των ενόπλων δυνάμεων και συγκεκριμένα και με αυτούς που βρίσκονται στα ανατολικά της Ουκρανίας, πολλές φορές ακούσαμε ότι υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις τις οποίες θέτει πλέον η Ρωσία σε σχέση με τους άμεσους γείτονές της αρχής γενομένης από την Αρκτική, φτάνοντας μέχρι το Καλίνιγκρα, το Κουλέβιετς, όπου βλέπουμε πλέον ότι υπάρχουν στρατιωτικές ικανότητες που χρησιμοποιούν ακόμα και πυρηνικά όπλα, πυρηνικές κεφαλές. Αυτά είναι τα τελευταία νέα τουλάχιστον τα οποία μας φτάνουν και βέβαια υπάρχουν και πολλές άλλες στρατιωτικές προκλήσεις, πολύ πιο ανατολικά όπως η προσάρτηση της Κρυμαίας, οι στρατιωτικές επιθέσεις στην Ανατολική Ουκρανία, καθώς επίσης και η στρατιωτική ανάπτυξη της Ρωσίας, ακόμα και στην περιοχή της Μεσογείου, μέσω ασκήσεων. Ο θύλακας λοιπόν του Καλίνιγκραντ είναι καθοριστική σημασίας σε αυτό το γεωπολιτικό, απειλητικό περιβάλλον το οποίο αναδύεται όλο και περισσότερο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι οι εξελίξεις σε αυτή την περιοχή. Εγώ Προέρχομαι από το της Πολωνίας, εκεί μεγάλωσα, εκεί ζουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Και θυμάμαι ότι πριν από μερικά χρόνια, ορισμένοι λέγανε ότι ε, αυτή η απειλή της στρατικοποίησης ε, της περιοχής δεν υφίσταται πλέον. Και πραγματικά είχα αποθαρρυνθεί τότε και πραγματικά μπορώ να σας πω ότι μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας έχουμε και στη δική μου την περιοχή περαιτέρω πλέον εξελίξεις, τις οποίες δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε πριν από μερικά χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, περιμένουμε να γίνει και ο επόμενος γύρος συνομιλιών στα πλαίσια του ΝΑΤΟ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Φαντάζομαι ότι ο κύριος ε, Μπερνιέ θα αναφερθεί σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν μέχρι τότε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για τις προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας που έχουμε στην περιοχή του Καλίνιγκραντ. Γι' αυτό το λόγο δώσαμε ε, ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα αυτό της ημερήσιας διάταξης. Έχετε το λόγο. Μεγάλη μου τιμή να σας παρουσιάσουμε τις δικές μας απόψεις της δικές μας υπηρεσίες του Υπουργείου Αμήνης για την ε, περιοχή αυτή. πρώτα πρώτα να σας ευχαριστήσουμε γιατί αναδείξατε αυτό το θέμα και το θέσατε προς συζήτηση εδώ στην ε, Επιτροπή Αμήνας και Ασφάλειας. Είμαι θα ότι η κατάσταση επιδεινώνεται στην περιοχή της Βαλτικής. Και όλα αυτά εντάσσονται στι εξελίξεις ε, για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας στην Ευρώπη. Τώρα για να δούμε μια σφαιρικότερη ε, εικόνα των ε, απειλών της βάρος της ασφαλείας στην Ευρώπη, πριν δούμε συγκεκριμένα τα της Βαλτικής να αρχίσω, λέγοντάς σας ότι υπάρχουν κάποιοι ευρύτεροι στόχοι της ρωσικής ηγεσίας όσον αφορά την Ευρώπη τουλάχιστον ε, τα τελευταία 10 χρόνια φαίνεται ότι στρατηγικός στόχος της Ρωσίας είναι να υπονομεύσει την κατάσταση της ε, ασφαλείας μετά την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Να υποκαταστήσει τα όσα ασχύουν με κάτι άλλο. Άρα πρόκειται εδώ για έναν κίνδυνο αυτής της αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Γι' αυτό και συνέχεια είναι αντίθετη στην επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς και με κάθε μέσο προσπαθούν να σπάσουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Θέλουν να δημιουργήσουν ή να παροξύνουν τις προστριβές, τις συγκρούσεις, επικαλούμενοι τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό και είχαμε την προσάρτηση της Κρυμαίας και τα όσα έγιναν στην Ανατολική Ουκρανία. Οπότε έχουμε τώρα μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού των όπλων δυνάμεων έχουμε κάποιες ε, ασκήσεις τεωρητικές χωρίς προηγουμένη προειδοποίηση. Όλα αυτά εντάσσονται στην τάση αυτή της ε, στρατηγικής της Ρωσίας. Βάση είναι η στρατηγική ισχύς, αλλά και η προθυμία να μετέρθουν την στρατηγική αυτή ισχύ και να επιβάλλουν τόσο θέλουν. Έχει έρθει το ΝΑΤΟ δυνάμεις, αλλά αυτό το λίγο που να κάνουν ότι στα ανατολικά σύνορα της, ε, των χωρών του ΝΑΤΟ θέλουν να έχουν ε, την ισορροπία δυνάμεων υπέρ τους. Οπότε έτσι να ε, μπορούν να αποσπάσουν ωφέλιο βραχυπρόθεσμα. Επίσης, δείχνουν την ισχύ τους. Δεν θέλουν όμως να υπάρξει απευθεία σύγκρουση με ισχυρούς αντιπάλους και εφευρετικούς, το μπορούμε να πούμε. Το 2008 στην Ουκρανία, το 2014 και στη Συρία φέτος είδαμε τι κάνει η Ρωσία. Δοκιμάζει την αντοχή, τη δύναμη των αντιπάλων. Έχουν πολλά μέσα. Στρατιωτική διπλωματία, κατασκοπία, προπαγάνδα, ε, διαχείριση της πολιτικής εξουσίας για τις κατοικούς καταστάσεις έχουν δηλαδή ευελιξία και την ικανότητα να επιχειρούν σε πολλά επίπεδα και σε πολλούς τομείς. και δε Βαλτική έχουμε κάποια κρίσιμα σημεία και εκεί έχει πετύχει μεγάλη συνέργεια η Ρωσία. Ο εξυγχρονισμός είπαμε, ιδίως όσον αφορά την δυτική περιοχή και έχουμε και επέκταση και παρέκταση των δυνατοτήτων τους. Έχουμε γυμνάσια στρατιωτικά και προκλητικές επιχειρήσεις. Όσον αφορά τώρα τον εξυγχρονισμό, ε, έχουμε επίσης κοντά σε αυτόν και αύξηση του στρατού, στρατικής ισχύω. Ξεκίνησε αυτό το 2015 σε αυτή την δυτική περιοχή. Πρόκειται για κάποιες μεταβολές οι οποίες μας παραπέμπουν σε εποχές ψυχρού πολέμου. Από τότε που άρχισε επομένω ε, αυτή η προσπάθεια αλλαγή το 2000 έχουμε δύο τάσεις όσον αφορά τις ε, μεταβολές στην κατάσταση εκεί. Πρώτα πρώτα η ενίσχυση των μονάδων αυτό που περνάνε τον εξοπλισμό και επίση τώρα έχουν νέε μονάδε εξυγχρονισμένε που είναι τοποθετημένες κοντά στα σύνορα με την Πολωνία οπότε έτσι υπάρχει μια σημαντική συγκέντρωση δυνάμεων και αυτό θα είναι χρήσιμο να θέλουν να κάνουν ε, κάποια επίθεση σε ένα περισσότερα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Τώρα επίση υπάρχει αυτό το πλάνο που ξεκίνησε το 2000 και έχουμε επομένω κάποιες μικρές ε, μονάδες οι οποίες τώρα έχουν καταργηθεί στην περιοχή τη Βαλτική. Παρ' όλα αυτά όμως το προσωπικό των μονάδων έχει αυξηθεί. Αυτό είναι Το 2009 η 25η τεραγμένη ημεραρχία πήγε κοντά στα σύνορα της Εστονίας. Το 2013 ανοίξανε πολύ κοντά στα λετωνικά σύνορα ένα στοτικό αεροδρόμιο. Και ανέπτυξαν και μια μεγάλη μονάδα, μια πτέρυγα μάχη τέλο πάντων με ελικόπτερα. Σε πάρα πολλέ μονάδε έγινε αναβάθμιση και στο Καλίνιγκραντ επίση έχουν άλλε δυνάμει και τώρα υπάρχουν καινούργια οχήματα μεταφοράς αρμάτων. Και στην Αγία Πετρούπολη έχουν 72 καινούργια άρματα και άλλα τεθροκισμένα οχήματα. Όλα αυτά είναι τακτικές μεταβολές καταρχήν, αλλά όλα μαζί εάν τα αφρίσετε σημαίνει αύξηση της συστατητικής ισχύω. Επομένως βλέπουμε ότι στην περιοχή της Βαλτικής έχουμε αύξηση της ρωσικής στρατηγικής παρουσίας. Όμως δεν πρόκειται μόνο για αυτό. Ε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα εκεί στην περιοχή της Βαλτικής πρόκειται για αυτή τη νέα ανάπτυξη και υπάρχει μια δύναμη αναστολής Επίσης ε, ε, εκμεταλλεύονται και την περιοχή της ε, Λευκορωσίας οπότε πρόκειται για μια απειλή παρόμοια αυτού του είδους οι στρατηγικές δυνατότητες αναπτύσσονται και σε άλλες περιοχές όπως τη Μαύρη Θάλασσα αλλά και την Συρία. Έχουν προχωρημένο σύστημα με πυράβλους S-400 στο Καλίνιγκρατ και στην Αγία Πετρούπολη. Και επίσης αυτά τα συστήματα ε, συνδυάζονται και με τα συστήματα που έχουν στην ε, Λευκορωσία. Οπότε είναι κοντά στην Ανατολική Πολωνία και έτσι ελέγχουν σχεδόν πάσα κίνηση στον ενέργειο χώρο αυτής της περιοχής. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι φαλιστικοί πύραυλοι μικρού βελνικού και μπορούν έτσι να στοχεύσουν κάθε στρατηγικό στόχο. Σιδηροδρόμους, ε, αεροδρόμια, στρατό, σιδηροδρόμους επίσης από τη Γερμανία μέχρι τη Φιλανδία και ταυτόχρονα ε, μπορούν επομένως να προστατευτούν σε πάρα πολύ μικρό χρόνο από αυτή την ε, άμυνα αέρος, εδάφος αέρος μόνο. Επίσης, τα αεροπλάνα μπορούν να βυστήσουν στην περιοχή του ΝΑΤΟ παρά τα συστήματα συναγερμού. Και υπάρχει αυτός ο anti-access factor, όπως ονομάζεται και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά μεταφορικά επομένως και έτσι για να απλουστεύσουμε μπορούμε να πούμε ότι εκεί υπάρχει αυτό το σύστημα που μπορεί, το σύστημα άμυνας που μπορεί να θεωρηθεί το ξύφος και η βαλιστική πύραυλη S400 ή ασπίδα. Από το 2007 έχουν αναβαθμίσει επίσης τον οπλισμό ε, και κατά θάλασσα. Έχουν τις που έχουν πυράβλους, μπορούν να χτυπήσουν ε, σε μεγάλη απόσταση και με ακρίβεια στόχου στην ξηρά. Αυτά δεν υπήρχαν πριν στη Βαλτική. Ακόμα και τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκαν οι δυνατότητες στην περιοχή. Και ανέπτυξαν στο Καλίνιγκραντ φρεγάτες με πυράβλους, κρούζ και άλλους μπορούν επομένω να χτυπήσουν ακόμα πιο μακριά στην Ευρώπη με αυτού. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν κινδύνους κλιμάκωσης. Είναι δύσκολο να χτυπηθούν σαν στόχοι οι ρωσικές δυνάμεις εκεί και είναι πάρα πολύ δύσκολο το ΝΑΤΟ να βοηθήσει και να ενισχύσει τους, ε, τα ανατολικά κράτη-μέλη. Επίσης δυσκολεύεται η στρατηγική επικοινωνία μεταξύ Πολωνίας και Βαλτικών χωρών. Συστηματικά λοιπόν αναβάθμιζαν τις δυνάμεις τους οι Ρώσοι, ούτως ώστε να έχουν ε, πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες να αναπτύξουν επιχειρησιακή δυνατότητα και έτσι τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση επιχειρήσεων έχουν το πάνω χέρι. και ελαφρά αεροσκάφη στην περιοχή εκεί που μπορούν αυτά να πλήξουν τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ εάν το ΝΑΤΟ να κάνει κάποιες μεταφορές. Επίσης μπορούν να χτυπήσουν σε όλη την περιοχή της Βαλτικής στόχους κατά ξέρα αν υπάρξει κάποια κρίση. Οπότε ακόμη και αν χρειάζεται μια τέτοια συγκέντρωση δυνάμεων για μια επίθεση σε Συρία και Γεωργία αλλά και Ουκρανία αποδεικνύει ότι μπορούν να αναπτύξουν δυνάμεις σε μεγάλες, σε μεγάλες αποστάσεις και γρήγορα. Μπορούν να τις υποστήριξουν επίσης πολύ καιρό. Και οι δυνάμεις στη δυτική περιοχή της ε, Βαλτικής επίσης μπορούν να ενισχυθούν από άλλα σημεία στη Ρωσία και με πρόφαση της ε, ασκήσεις στα γυμνάσια. Επομένως, αν υπάρξει κάποια ένοπλη αναμέτρηση στη Βαλτική, εάν το ΝΑΤΟ δεν προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση, δεν υπάρχουν πάρα πολλές ε, επιλογές, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε την κλιμάκωση και να αποφύγουμε το σενάριο του να κερδίσουν ε, κάποια εδάφη, κάποια σημεία οι Ρώσοι. Ε, οπότε έχουν αναπτύσσουν τις δραστηριότητες προκλητικές. Πληροφόρηση, ιδεολογικά, διπλωματικά, κάθε είδους προκλήσεις, αλλά οι επιχειρήσεις κυρίως θέλουν ούτως ώστε να παραπλανήσουν τι στρατιωτικές αρχές και τι πολιτικέ αρχές των άλλων χωρών. Έχουν και αποσταθεροποιητική προπαγάνδα, ούτως ώστε επίσης να δημιουργήσουν προβλήματα στις κοινωνίες. Έμεσα επομένως κινούνται και επίσης ε, ε, θέλουν, κάνουν κάποιους αποκλεισμούς, ε, ζώνες απαγόρευσης πτήσεων και επομένως αυτό είναι ο υβριδικός πόλεμος, το υβριδικό φαινόμενο. τις δε στρατιωτικές επιχειρήσεις υπάρχει το φαινόμενο ότι είναι ασαφής η διάκριση μεταξύ αυτού του υβριδικού πολέμου και του πραγματικού πολέμου. Υπάρχει επομένως αυτή η απειλή κατά της ευρωατλαντικής συνοχής. Οπότε αυτό το στρατιωτικό δόγμα ισχύει για πολλούς τομείς και μας δείχνει ότι δεν είναι μόνο κάτι θεωρητικό. Η παρουσία στην Βαλτική από στρατιωτικής αυξάνεται και δικαιολογεί τον προβληματισμό όλων των χωρών του ΝΑΤΟ. Και αυτές οι δυνατότητες AD όπως ονομάζονται είναι στρατηγική. Έτσι μπορούν να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για επίθεση πάσης κλίματος. Χρειάζεται επομένω μια μακρόπνοη στρατηγική αντιμετώπισης. Στη Βαρσοβή, σαν της κορυφής, το συζητήσαμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αν θέλετε να συζητήσουμε για να σας απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας αυτή. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Ντέιβις Πετραϊτής, ο οποίος εκπροσωπεί το Υπουργείο Άμυνας της ε, Λιθουανίας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω σήμερα εδώ. Δεν θα αναλώσω πάρα πολύ χρόνο στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων, θα περάσω στην στρατιωτική διάσταση των πραγμάτων και μάλιστα θα επαναλάβω εν μέρει αυτά τα οποία είπε Το πρώτο σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να συντοπίσουμε είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντε που επιφέρουν πλέον κάποιε αλλαγέ στην επικρατούσα κατάσταση στη Βαλτική. Βλέπουμε ότι οι Ρώσοι όλο και περισσότερο προχωρούν σε ενορχιστρωμένες στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις. Έχουν λοιπόν κάποιες νέες δυνάμεις, κάποιες νέες συμβατικές δυνάμεις, χρησιμοποιούν πολεμικά δόγματα μάχης και παράλληλα βλέπουμε ότι ένα από τα δόγματα αυτά προβλέπει ότι η Ρωσία θα έχει μια προσέγγιση οχυρού όπως λέγεται όσον αφορά την αμυντική της στρατηγική και το Καλίνιγκραντ αποτελεί μία από τις περιοχές αυτές. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μερικές φορές δίνει την εντύπωση ότι η Ρωσία ασχολείται μόνο με τη Δύση, ενώ στην πράξη υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι η Ρωσία δημιουργεί ανάλογες στρατιωτικές δυνατότητες και ικανότητες σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται. Υπάρχει δηλαδή ένα συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών αμυντικών δραστηριοτήτων της Ρωσίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι δημιουργούνται νέες στρατιωτικές δυνάμεις, εξοπλίζεται εκ νέου η Ρωσία και δημιουργεί νέα στρατιωτικά δόγματα. Στη γραφική αυτή παράσταση βλέπετε κάποια σημαντικά γεγονότα που καταδεικνύουν ότι όντω σημειώνει πολύ σημαντική στρατιωτική πρόοδο η Ρωσία. Βλέπετε τις αλλαγές που έχουν επέλθει μέχρι σήμερα, βλέπετε τις νέες δυνάμεις που έχουν δημιουργηθεί, τις λεγόμενες ήπιες δυνάμεις και στη συνέχεια τις λεγόμενες σκληρές δυνάμεις. Και βλέπετε ότι ακόμα και στην περιοχή του Καλίνιγκρατ και οι δύο κατηγορίες δυνάμεων είναι παρούσες. Και βλέπετε ότι εφαρμόζεται και περισσότερο το δόγμα του υβριδικού πολέμου. Ας επικεντρωθούμε τώρα στη στρατιωτική πτυχή των πραγμάτων. Βλέπετε για παράδειγμα εδώ κάποιες περιπτώσεις εξυγχρονισμού των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας. Στο πρώτο στάδιο, γιατί βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο, προσπαθούσαν να εξυγχρονίσουν τις υφιστάμενες δυνάμεις τους, να γίνουν σύγχρονες στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια νέων τακτικών στρατιωτικών δογμάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο, αποσταθεροποιούνται οι υπόλοιπε στρατιωτικέ διοικήσει των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, γιατί καλούνται τώρα να προσαρμοστούν στο νέο εξοπλισμό της Ρωσίας, που πολλές φορές ο δικό μας τελικά εξοπλισμός υστερεί. Όσον αφορά τα στρατιωτικά δόγματα τα οποία χρησιμοποιεί η Ρωσία, ένα από αυτά το αναφέραμε ήδη, πρόκειται για το A2AD, δηλαδή αυτό το δόγμα απαγόρευση πρόσβασης και περιορισμού της πρόσβασης. Υπάρχει όμως και ένα άλλο δόγμα που έχει να κάνει με τα όπλα ακριβίας μεγάλου βεληνικούς που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, αλλά και σε τακτικό στρατιωτικό επίπεδο χρησιμοποιούνται κάποιες νέες μέθοδοι. Να σας δώσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Για παράδειγμα, ηλεκτρονική πλέον διεξαγωγή πολέμου, μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τη Ρωσία, Βλέπετε επίσης ότι έχουμε νέες υβριδικές προσεγγίσεις, όπως για παράδειγμα χρησιμοποίηση πλέον ειδικών δυνάμεων, που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο κοντά στα ευρωπαϊκά σύνορα και παράλληλα βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι χρησιμοποιούνται νέες οπτικές μέθοδοι στα όπλα τα οποία χρησιμοποιεί η Ρωσία και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερες επιζήμες επιπτώσεις στις δικές μας τις δυνάμεις. Όλα αυτά τα φαινόμενα τα βλέπουμε να αναδύονται όλο και περισσότερο στο Καλίνιγκραντ. Ήδη επί του παρόντος στο Καλίνιγκραντ έχουμε στρατιωτικές δομές οι οποίες είναι παγιωμένες και οι οποίες υφίστανται, όπως σας είπα, ήδη από σήμερα. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες ταξιαρχίες οι οποίες εξοπλίζονται όλο και περισσότερο. Φαντάζομαι ότι θα διαβάσατε ότι η Ρωσία θα αυξήσει τα τάγματα αναγνώριση τα οποία έχει στην περιοχή. Χρησιμοποιούνται λοιπόν όλο και περισσότερο νέα στρατιωτικά δόγματα πάρα πολύ κοντά στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερθήκαμε επίση στο δόγμα A2AD, το οποίο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Το Καλίνιγκρατ είναι ένα μόνο, μία μόνο από τι τέσσερι περιοχέ όπου χρησιμοποιείται το δόγμα αυτό. Η Ρωσία προσπαθεί να επιβάλλει το δόγμα αυτό απαγόρευση πρόσβαση και στην Κρυμαία στην Χερσόνησο Κόλα, στις Κουρίλες Νήσους και στο Καλίνιγκραντ. Αν εξετάσουμε εκ του συνεγγιστή κάουνε στην πραγματικότητα οι Ρώσοι, βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής το Καλίνιγκραντ αποτελούσε η τελευταία προτεραιότητα της Ρωσίας και μόνο τελικά τους τελευταίους μήνες η Ρωσία άρχισε να αναβαθμίζει αυτή την προτεραιότητα καθότι κατάφερε να καλύψει τις τρεις άλλες προτεραιότητες οι οποίες προηγούνταν. Πρόσφατα για παράδειγμα, είδαμε ότι υπήρχαν όλο και περισσότερες ε, μετακινήσεις αμυντικών συστημάτων προς το Καλίνιγκραντ, πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι όντως η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα οχυρό γύρω από το Καλίνιγκραντ. Βλέπετε εδώ πέρα μια γραφική παράσταση για το τι μπορεί να καλύψει γεωγραφικά το νεο αυτοδογμα δόγμα A2AD, απαγόρευσης πρόσβασης ή περιορισμού πρόσβασης. Βλέπετε ότι υπάρχει ήδη μια αμυντική περιοχή προστασία που είχε δημιουργηθεί από του Ρώσου. Βλέπετε επίση ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα οχήματα Ισκαντέρ, το τακτικό αυτοσύστημα βαλιστικών πυράβλων. Όλο και περισσότερο πλικά τέτοια συστήματα, αλλά και νέες μονάδες της ε, πολεμικής αεροπορίας χρησιμοποιούνται στην περιοχή αυτή, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η αντιπυραυλική ασπίδα. Αν δούμε επίση τι κάνουν στι παράκτε περιοχέ οι Ρώσοι, βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι οι Ρώσοι έχουν ήδη αρχίσει να κινούν προ τι παράκτε περιοχέ ένα νέο σύστημα χρησιμοποίηση πυράβλων κατά πλοίων. Είμαστε σίγουροι ότι θα αρχίζουν να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν τα, συστήματα αυτά όλο και περισσότερο. Πιστεύω λοιπόν ότι πολύ σύντομα οι Ρώσοι θα δημιουργήσουν ένα πολύ ισχυρό οχυρό, το οποίο θα βρίσκεται πραγματικά πάρα πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουν στα πλαίσια του συστήματος αυτού μια πολύ ισχυρή στρατιωτική συνιστόσα η οποία θα μπορέσει να χτυπήσει πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων όμορων χωρών. Βλέπουμε επίση ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ένα πολύ κεντρικό σύστημα στρατιωτική διοίκηση. Εδώ και ένα χρόνο δημιούργησαν ένα εθνικό κρατικό κέντρο αμυντικού συντονισμού. Όλο και περισσότερο λοιπόν η ρωσια χρησιμοποιει ενα πολυ κεντρικο συστημα στρατιωτικης διοικησης εδω και ενα χρονο δημιουργησαν μπορεί να συντονίζει όλες τις στρατιωτικέ τη δραστηριότητε τόσο στο Καλίνιγκρα όσο και σε άλλες περιοχές. Ακούσαμε ήδη ότι έχουν σημαντικέ στρατιωτικέ ικανότητε, ότι προσπαθούν να κινήσουν συγκεκριμένε στρατιωτικέ μονάδε σε πολλέ περιοχέ του κόσμου, προειδοποιώντα ουσιαστικά την τελευταία στιγμή. Και βλέπετε ότι το κέντρο αυτό αμυντικού συντονισμού μπορεί πραγματικά να συντονίζει όλε αυτέ τι διαφορετικέ στρατιωτικέ δραστηριότητε σε πάρα πολλέ περιοχέ του κόσμου. Και αναφέρομαι εδώ πέρα μόνο στην αμυντική πλευρά των πραγμάτων. Βλέπετε εδώ ότι η περιοχή του Καλίνιγκρατ είναι στα κάτω αριστερά της γραφικής αυτής παράστασης. Βλέπετε δηλαδή ότι ήδη το Καλίνιγκρατ έχει από τακτικής πλευράς συμπεριληφθεί στο κέντρο αυτού συντονισμού της ε, Ρωσίας. Μαζί με άλλες περιοχές βέβαια που περιλαμβάνονται εκεί και δεν χρειάστηκε να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να το πετύχει αυτό η Ρωσία. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε ότι τα όσα συμβαίνουν στον Καλίνιγκραντ δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ε, μεμονωμένες δραστηριότητες της Ρωσίας, αλλά εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο στρατιωτικό της Ρωσίας, προκειμένου να καταφέρει να αυξήσει σε διάφορα μέρη του πλανήτη τη στρατιωτική της παρουσία. Βλέπετε εδώ το σύνολο των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Ρωσίας όχι μόνο στο Καλίνιγκρατ αλλά και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, προσπάθησαν να δημιουργήσουν κάποιες νέες ταξιαρχίες. Ταξιαρχίες που έχουμε στο Καλίνιγκρατ τις βλέπουμε και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Μόλις άρχισαν να εφαρμόζουν τον δόγμα των κοινών στρατιωτικών δυνατοτήτων, άρχισαν να μεταφέρουν στο Καλίνιγκραντ τα αμυντικά συστήματα Ισκαντέρ και φαίνεται ότι θα βρίσκονται πλέον μόνιμα σε ένα καθεστώς μόνιμης εγκατάστασης στα συστήματα αυτά στο Καλίνιγκρατ. Όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι ε, από στρατοτικής τουλάχιστον πλευράς, από πλευρά στρατοτικών ικανοτήτων, θα πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε πάρα πολύ στη σοβαρά υπόψη την παρουσία των Ρώσων στο Καλίνιγκραντ. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ε, η στρατιωτική αυτή δραστηριότητα αποτελεί απλώς ένα εργαλείο της πολιτικής βούλησης, της πολιτικής διοίκησης της Ρωσίας. Βλέπετε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν είπε ορισμένα πράγματα σε ένα φόρουμ το οποίο έλαβε χώρα πρόσφατα τον Οκτώβριο. Η χώρα αυτή μας λέει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ζητήσει τη δική μας την άδεια προκειμένου να κινηθεί στρατοτικά σε συγκεκριμένες περιοχές. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να λάβει υπόψη της τις δικές μας τις ανάγκες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να είμαι σε θέση να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πετράητης. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπερνιέ. θα ήθελα. Αλλά προηγουμένω θα ήθελα να σας ε, ζητήσω να σηκώσετε το χέρι σας αν θέλετε να πάρετε το λόγο στη συνέχεια. Κύριε Μπερνιέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερως. Σας ευχαριστώ επίσης ε, τους ε, άλλους ομιλητές για τις πληροφορίες αυτές που είναι πολύ, των insiders που είναι πολύ χρήσιμες για μας στην ανάπτυξη της δικής μας πολιτικής. Εντάχει, θα ήθελα να πω τα εξή. Όπως είπε ο άλλος συμμιλητής, το στοιχείο στρατηγικοποίησης στο Καλίνιγκρεντ θα πρέπει να τοποθετηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας της ε, Ρωσίας, ε, της προβολής μιας ε, ισχύω προς τα έξω την ε, προθυμία άσκησης ε, δύναμης κλπ. Το άλλο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό είναι να έχουμε κατά νου την ε, στρατηγική σημασία της περιοχής της Βαλτικής. Και πρόκειται ακριβώς για την περιοχή του κόσμου που η Ρωσία έχει σύνορα τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με τον ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν Εκεί είναι, ε, η έννοια της ζώνης επιρροής της Ρωσίας ε, καθώς και τα τροτά σημεία της Ρωσίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για μια περιοχή όπου υπάρχει μια κρίσιμη υποδομή για τις, ε, τα ευρωπαϊκά κράτη και τους συμμάχους Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα περιβάλλον που ασκούνται διάφορες πιέσεις. Η στατιστική σημασία της περιοχής του Καλίνιγκρατ μας ε, υποχρεώνει τους ε, ε, Ρώσους να αναπτύξουν τις δυνάμεις τους και να ασκήσουν πίεση στους μάχους τους και στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης είναι μια Επίσης ε, ε, θεωρώ ότι η άμυνα του Βόρειου Στόλου της ε, Ρωσίας δράζεται εκεί κάτι εξαιρετικά σημαντικό από την προοπτική της Ρωσίας. Όσον αφορά τη στρατηγικοποίηση του ιδίου του Καλίνιγκραντ, ε, ε, σε σχέση με την αμυντική πολιτική του ΝΑΤΟ, θα ήθελα να πω ότι είναι τμήμα ενός ευρύτερου πλαισίου, όπως ήδη έχει αναφερθεί, που αφορά ένα μέτωπο άσκηση στρατιωτικής δραστηριότητας από την Βαλτική έως την Μεσόγειο. Όλα λοιπόν τα οποία συμπεριλαμβάνουν ακριβώς την εγκύτητα των συμμάχων συμπεριλαμβάνοντας τα θέματα της προσάρτησης της ε, Κρυμαίας και τις επιχειρήσεις ε, σε σχέση με τη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά τη δική μας προοπτική του ΝΑΤΟ, η παρουσία των στρατικών δυνάμεων ε, της Ρωσίας δεν είναι το πρόβλημα. Το δικό μας θέμα είναι να αναπτύξουμε τις δικές μας δυνάμεις ε, στο πλαίσιο ακριβώς της ε, προσπάθειας της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Οι στρατιωτικές δυνατότητες περιγράφησαν πολύ καλά από τους δύο συναδέλφους και ε, σε σχέση με τα πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνικού, τους πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους και όλα αυτά συγκεντρώνονται ε, στην συνολική, στο συνολικό δυναμικό των ρωσικών δυνάμεων. Πρόκειται για αμυντικές δυνάμεις που μπορούν να έχουν επιθετική εμβέλεια σε σχέση με το, την επικράτεια του, των συμμάχων. Η ε, κίνδυνη ε, εδώ στο Καλίνιγκρατ είναι να γίνει ένα είδος πλατφόρμας de facto ε, σε σχέση με τους ε, συμμάχους όσον αφορά την ε, επίσης να η ελεύθερη ναυσιπλοεία και υπάρχουν αναρίθμητα παραδείγματα σε άλλες χώρες που δίνουν έναυσμα για ανησυχίες. Και αυτού του είδους αρσιδιότητες στο ευρύτερο πλαίσιο το οποίο είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια ήταν λόγος για λήψη αποφάσεων εκ μέρους του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα στη Σύνοδο Κορυφής που έγινε το 2014, ε, όπου εκπονήθηκε ένα πρόγραμμα δράσης και έγινε και μια συνάντηση τον τελευταίο Ιούλιο όπου δόθηκε έμφαση σε θέματα άμυνας. Ε, από, από την προπτική την οπτική γωνία του ΝΑΤΟ, τα μέτρα τα οποία λάβαμε είναι αμυντικής ε, φύσεως ε, και είναι συνεπή με τις ε, δεσμεύσεις μας και καταδεικνύουν ακριβώς την προσπάθειά μας να προβούμε σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική η οποία να βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες. Και βεβαίως αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό για μας. Αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό επίσης να δούμε είναι ότι στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δικής μας θέσης έχουμε την πόρτα ανοιχτή για, ένα, για κίνηση διαλόγου με τους Ρώσους και την ανάληψη δεσμεύσεων. Ο στόχος είναι βεβαίως να υπάρχει μια διαφάνεια και μείωση των κινδύνων. Και αυτή είναι μια ε, σύνθετη προσπάθεια, αλλά που είναι σημαντική, καθοριστική για μα. Δύο εβδομάδε μετά την Σύνοδο Κορυφή στη Βαρσοβία είχαμε μια συνάντηση ε, ΝΑΤΟ και Ρωσία, όπου παρουσιάσαμε τα μέλη μας ε, στην Ρωσία και επίσης επισημάναμε την ανάγκη η Ρωσία να παρουσιάσει με ένα διαφανή τρόπο τη δική της ε, θέση και το, το πλαίσιο των δικών της ασκήσεων, όπως κάναμε και εμείς προηγουμένως από τη δική μας πλευρά. Ένα ε, σημαντικό σημείο όσον αφορά τη δική μας θέση στο πλαίσιο του Καλίνιγκρατ, στο πλαίσιο των ζητημάτων ασφαλείας που έχουμε στην περιοχή της Βαλτικής, είναι μια από τις πιο συμβολικές αποφάσεις οι οποίες ε, λήφθησαν στην Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας, δηλαδή την ενίσχυση της παρουσίας ε, του ΝΑΤΟ στην ε, Βαλτική και στην Πολωνία. Και πρόκειται για μια ταπεινή παρουσία ε, εκ μέρους μας. Το πρόβλημα δεν είναι δεν είναι να αναπτύξουμε πλήρως τις δικές μας δυνάμεις σε σχέση με τη Ρωσία, ε, εμείς το, θέμα είναι ένα περιφερειακό σενάριο. Ε, ωστόσο υπάρχει και ένα σενάριο υβριδικής φύσης. Δηλαδή είναι δύσκολο να υπάρξει επιμερισμός ευθυνών εδώ δηλαδή η δική μας διαδικασία λήψη αποφάσεων είναι πιο σύνθετη και πιο δύσκολη. Χάνουμε χρόνο, χάνουμε πρωτοβουλίες και αυτό ακριβώ θέλουμε, περιθώριο ανάπτυξης πρωτοβουλειών και γι' αυτό θέλουμε να αποφύγουμε και γι' αυτό είπαμε στη Βαρσοβία ότι θα πρέπει να ε, έχουμε δυνατότητα να άρουμε όλες αυτές τις αμφισημίες, ε, να υπάρξει μια ε, δυνατότητα διευκόλυνσης της λήψης πολιτικών αποφάσεων. Από την δική μας οπτική γωνία είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν εκφράζουμε, δεν εκτοξεύουμε απειλές προς καμία πλευρά, ούτε τη Ρωσία. Γι' αυτό έχουμε μια διαφανή θέση και έχουμε μια διαφάνεια σαν ασφορά τη δική μας ανάλυση της κατάστασης ασφαλείας στο Καλίνιγκρατ και ευρύτερα στην ε, περιοχή της Βαλτικής. Σημαντικά στοιχεία είναι οι γενικότερες επιπτώσεις εδώ. Η πρώτη επίπτωση είναι το ενδιαφέρον πολλών εταίρων, Σουηδίας και Φιλανδίας ιδιαίτερως, να συζητήσουν ε, θέματα ασφαλείας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ με ένα ανοιχτό και διαφανή τρόπο, με όλους τους συμμάχους. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα δείγμα της ποιότητας της δικής μας ανάλυσης ε, για την περιοχή και μια άλλη επίπτωση είναι η συνειδητοποίηση της σημασίας της ανταλλαγής ε, πληροφοριών μεταξύ των συμμάχων. Επίσης η έννοια του συντονισμού, η έννοια της ε, παρουσίασης των στρατηγικών, πώς προσλαμβάνεται από τους άλλους και πώς ε, μπορούμε ε, να αναπτύξουμε τις δικές μας αντιδράσεις. Ένα άλλο θέμα. Ε, πολλές από τις ασκήσεις των Ρώσων τις γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες άλλες ασκήσεις πέρα από αυτές που προαναγγέλουν. Ε, το πώς ε, αντιδρούμε εμείς ε, είναι σημαντικό εδώ. Επίσης, το θέμα της προετοιμασίας σε πολιτικό, των πολιτών και αυτό είναι σημαντικό. Το ζήτημα λοιπόν της θετικοποίησης της ζώνης του Καλίνιγκρατ είναι σημαντικό, είναι σύνθετο ε, λόγω της στρατηγικής σημασίας της περιοχής, όπου εδώ έχουμε κάποιες ξεκάθαρες ε, απαντήσεις. Θέλουμε να αυξήσουμε την ασφάλεια για την Ευρώπη, αλλά βεβαίως ε, δεν λύνεται τόσο απλά το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σε ενημερώσω πριν ξεκινήσουμε τώρα την γενικότερη συζήτηση για το θέμα αυτό, ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τίναντ με πυρογνώμονες ε, του ΝΑΤΟ και Γερμανών στρατηγών οι οποίοι συζήτησαν με θέματα γενικής φύσεως τη δέσμευση του ΝΑΤΟ στην ε, ανατολική και νότια πλευρά ε, στο, του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο ακριβώς των προκλήσεων. Και η άποψη που κυριάρχησε ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ε, πολυμερής ε, προσέγγιση η οποία ε, μπορεί να υπερκεβεράσει τις προσπάθειες των Ρώσων. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε αφελείς και μάλλον θα πρέπει να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αναλαμβάνουμε δράση και δεσμευόμαστε σε πολλούς τομείς προκειμένου να έχουμε μια επαρκή μόχλευση σε σχέση με τη Ρωσία, όχι μόνο στο στρατιωτικό επίπεδο, στη στρατιωτική σφαίρα, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς, γιατί ε, μπορέσαμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα ιδιαίτερα από την κατάσταση ιδιαίτερα το 2007 και το 2008 με την, τον πόλεμο στη Γεωργία και στη συνέχεια βεβαίως με την επίθεση και της Ουκρανίας και, στην Ουκρανία και την προσάρτηση της Κρυμαίας. Και νομίζω ότι παρόλα αυτά θα πρέπει να συνδυάσουμε πολλά όπλα και εργαλεία, στρατιωτικά και πολιτικά, ούτω ώστε να μπορέσουμε αποτελεσματικά να αποτρέψουμε την Ρωσία. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Γιαρομίλη Στρατσίνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι φορέστε, παρακαλώ πολύ τα ακουστικά σα. Θα μιλήσω τσέχικα. Δύο ερωτήσει θέλω να κάνω. Η πρώτη απευθύνεται στον κύριο Γκαμπριέλ Ντανιέ. Ακούσαμε κάτι για Green Man, αυτό είπατε. Το άρθρο 5 της συνθήκης μας θα μπορούσε να συσχετιστεί με τη λειτουργία αυτού του Green Man σε οποιαδήποτε χώρα βρίσκεται κοντά στο Καλίνιγκραντ. Δεύτερον, απευθύνομαι στον αξιωματούχο από την Λουθωανία και στον αξιωματούχο από την Πολωνία όσον αφορά τους πυράβλους αυτούς ε, Ισκαντέρ που τους βλέπουμε πλέον εγκατεστημένους στην περιοχή του Καλίνιγκραντ. Δεν προκαλεί εντύπωση ανησυχία που εξέφρασε η πρόεδρος, διότι οι πύραυλοι αυτοί οι Σκαντέρ είναι πύραυλοι που έχουν εμβέλεια 500 χιλιόμετρων. Θα μπορούσαν να πληγούν όμως ακόμα και οι κάτοικοι της Βαρσοβίας. Το βεληνικές των πυράβλων αυτών φτάνει μέχρι εκεί σας υπενθυμίζω ότι όταν βρισκόταν η Τσεχοσλοβακία υπό την ρωσική κατοχή, υπό την κατοχή των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, οι Σοβιετικοί τότε διατείνονταν ότι ε, ουδέποτε είχαν εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στην επικράτεια της πρώην Τσεχοσλοβακίας και κατά πάσα πιθανότητα την ίδια δήλωση κάνουν τώρα και για το Καλίνιγκρατ. Εσείς γνωρίζετε αν τυχόν υπάρχουν τελικά πυρηνικά όπλα στην επικράτη του Καλίνιγκραντ σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν παρόν κατά την παρουσίαση των πρώτων ομιλητών. Λυπάμαι πραγματικά που η Ρωσία επέλεξε τελικά να προχωρήσει σε μια στρατιωτικοποίηση της περιοχής της Βαλτικής, και ασκεί κατά αυτόν τον τρόπο πίεση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στη Βαλτική. Θυμάμαι τη δεκαετία του 90 τα πράγματα ήταν εντελώ διαφορετικά. Υποτίθεται ότι η περιοχή του Καλίνιγκρατ θα ήταν μια ελεύθερη ζώνη εμπορικών συναλλαγών, ότι μπορεί ακόμα και να εντασσόταν στην εσωτερική αγορά, στην ενιαία αγορά. Βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν πάρει εντελώ διαφορετική τροπή τώρα. Βλέπουμε ότι η Ρωσία αποφάσισε να δείξει δημιουργική στάση με εντελώ διαφορετικό τρόπο όμως και θεωρώ ότι αυτό είναι επονίδιστο. Επονίδιστο ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο στη γενέτειρα του Εμμάνιουελ Κάντ. Φαντάζομαι ότι πριν από 200 χρόνια θα είχε άλλα πράγματα να πει αν έβλεπε πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση. Τώρα, ας περάσουμε στο ζήτημα της στρατιωτικοποίησης. Αυτή μπορεί να συμβεί και μέσω χερσαίων δυνάμεων, έτσι δεν είναι. Και τι θα συμβεί με τη Λιθουανία τι είδους συμφωνίας έχει η Λιθουανία με τη Ρωσία όσον αφορά τις μεταφορές, τις σιδηροδρομικές και δικές μεταφορές. Θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις συμφωνίες αυτές η Ρωσία για την ανάπτυξη των χερσαίων της δυνάμεων. Ελπίζω ότι στη δική μας, στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, ελπίζω ότι πραγματικά έχουμε εξετάσει όλες τις δυνατότητες μεταφοράς και διαμετακόμισης και ελπίζω ότι από στρατιωτική πλευρά η διάβλη αυτή είναι προστατευμένη, προκειμένου προφανώ να αποτρέψουμε τέτοιου είδου στρατιωτικές κινήσεις και μεταφορές. Κάτι ακόμα. Στο παρελθόν, η Ρωσία είχε προχωρήσει σε τέτοιες διευθετήσεις ε, στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ε, προβλεπόταν ότι ε, θα υπήρχαν τα κατάλληλα συστήματα προστασίας και από τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή εσείς στην Πολωνία, στη Ανθουανία, χρησιμοποιείτε συστήματα παρακολούθησης και επιτήρησης προκειμένου να μπορείτε να βλέπετε πραγματικά τι γίνεται από την άλλη πλευρά των συνόρων ή εξαρτάστε μόνο από τα δορυφορικά συστήματα επιτήρησης του ΝΑΤΟ. Και τι κάνετε όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης. Επίσης, ε, έχετε καλέσει παρατηρητές ε, όσον αφορά τις στρατιωτικες αυτες αυτές εξελίξεις από άλλα κράτη-μέλη. Πώς σχεδιάζετε ακριβώς να αντιδράσετε στο μέλλον. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Αν κάνω λάθος διορθώστε με, αλλά θεωρώ ότι η Ρωσία άρχισε να στρατιοκοπεί την περιοχή της Βαλτικής για δεύτερη φορά, ότι αυτό είχε συμβεί και στο παρελθόν. Μπορεί να κάνω και λάθος. Νομίζω ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να εξετάζουμε τη στάση της Ρωσίας στην περιοχή. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο και θα μπορούσαμε να τη συγκρίνουμε με το επίπεδο των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας. Εν γέννη θεωρείται ότι το ΝΑΤΟ είναι πολύ πιο ισχυρό στρατιωτικά, αλλά έχει και ένα αδύναμο σημείο, ένα αδύναμο κρίκο. Το ότι αρχίζει σιγά σιγά και επηρεάζεται από την ε, κατάσταση στη Ρωσία. Ο κύριο Παχόλσκι, για παράδειγμα, αναφέρθηκε στο όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στι χερσαίε δυνάμει τη Ρωσία και πώ αυτά επηρεάζουν τελικά τι στρατιωτικέ ικανότητε του ΝΑΤΟ. Αναφορέ γίνουν επίση στο πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία τη Ρωσία και είπατε ότι στη Βαλτική θάλασσα χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή δύο κορβέτε τελευταία τεχνολογία, οι οποίε είχαν χρησιμοποιηθεί από τη Ρωσία στη Συρία και ο, οι οποίες είναι πολύ πιο ισχυρές ακόμα και από τα συστήματα Ισκάντερ. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι ανησυχία πλέον. Όλοι παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς αυτές τις εξελίξεις, όλοι διαπιστώνουμε και αναλύουμε τις κινήσεις της Ρωσίας, προσπαθούμε να δούμε τι κάνει το ΝΑΤΟ, και πώς η αντίδραση του ΝΑΤΟ σχετίζεται τελικά με τις κινήσεις της Ρωσίας. ένα δύο πράγματα όμως μου κάνουν εντύπωση. Πρώτον, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις γενικότερα είναι ιδιαίτερα επαγγελματικές, χρησιμοποιούν επαγγελματίες οπλίτες και όχι τόσο πολύ στρατευμένους πολίτες. Βλέπουμε επίσης ότι οι στρατιωτικές ικανότητές τους όλο και αυξάνονται. Όχι μόνο έχουν πλέον τη δυνατότητα γρήγορης ανάπτυξης των δυνάμεών τους, αλλά μπορούν να αντιδράσουν πολύ γρήγορα σε αναπάντεχες επιθέσεις. Αυτό το είδαμε συγκεκριμένα και στη Συρία και στην Κρυμαία. Δεν είμαστε πάντα σε θέση βέβαια να προβλέψουμε ή να εντοπίσουμε τέτοιες επιχειρήσεις της Ρωσίας. Το πρόβλημα λοιπόν έγκυται στο εξής καλούμεθα εμείς να αντιδράσουμε σε αυτές τις νέες εξελίξεις. Και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Αν πραγματικά θέλετε να αντιδράσετε από στρατικής πλευράς, τότε αναγκαστικά δεν γίνεται παρά να περιοριστείτε σε κάποιες συμβολικές κινήσεις. Από στρατικής πλευράς, ουσιαστικά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε κάποιες χιλιάδες στρατιώτες 5.000 για παράδειγμα ή ακόμα και λιγότερους πιο κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αντισταθμίσει την τεράστια στρατιωτική δύναμη της Ρωσίας. Θεωρώ ότι αν κάνουμε τέτοιες μεταφορές στρατιωτικού προσωπικού, η κίνησή μας αυτή θα είναι καθαρά συμβολική. Μπορούμε να αντιδράσουμε με τρόπο διτό. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε τις δραστηριότητες ε, του ΝΑΤΟ στο σύνολό του και από την άλλη έχουμε τις μεμονωμένες δραστηριότητες των κρατών μελών. Και πραγματικά έχω μείνει έκπληκτος, γιατί ε, ανάμεσα στα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη έχουμε ορισμένα τα οποία δεν θέλουν να ενισχύσουν τις στρατικές τους δυνάμεις και τις στρατικές τους προσπάθειες. Εγώ κατάγομαι από την Πολωνία, η οποία αναγνωρίζει πλέον τη σοβαρότητα της κατάστασης και αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι οι αμυντικές μας δαπάνες είναι το 2% του ΑΕΠ μας. Άλλες όμως χώρες δεν επιθυμούν να δαπανίσουν πάνω από το 1% του ΑΕΠ τους και πολλές φορές δεν φτάνουν καν σε αυτό το ποσοστό χρηματοδότησης του αμυντικού κλάδου. Νομίζω ότι ως μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να μιλούμε ανοιχτά για το ζήτημα αυτό και προτού προβάλλουμε περισσότερες προσδοκίες ή απαιτήσει στο ΝΑΤΟ, ας δούμε καλύτερα εμείς τι κάνουμε στα δικά μας τα κράτη, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας περάσω και σε κάποια άλλα ζητήματα τώρα. Ακούσαμε ότι αναδύονται πάρα πολλές απειλές. Μία από αυτές σχετίζεται με το ότι ε, δεν έχουμε εμεί αντιπυραυλικά συστήματα δεν επαρκούν αυτά τα οποία υπάρχουν και δεν γίνονται επενδύσεις αυτή τη στιγμή, ακόμα και να αρχίσουν οι επενδύσεις ήταν ιδιαίτερα δαπανηρές και χρονοβόρες. Με τους υφιστάμενους λοιπόν πόρους και τις υφιστάμενες ελλείψεις μας, μήπως θα ήταν καλύτερα να μεταφέραμε κάποιες στρατιωτικές μονάδες, για παράδειγμα τρεις-τέσσερις ταξιαρχίες Patriot στην περιοχή αυτή, θα ήταν καλύτερα να τις μεταφέραμε εκεί στην περιοχή δηλαδή γύρω από το Καλίνιγκρατ. Επίσης, τα, τα προγράμματα κατάρτισης τα οποία έχουμε δεν επαρκούν. Ο κύριος Κέλαμ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ για την ενημέρωση. Είναι ρεαλιστική η ενημέρωση. Και όχι μόνο οι πολίτες αλλά και εμείς οι πολιτικοί αισθανόμαστε ανήσυχοι. Το Καλίνιγκραντ έχει καταστεί το σύμβολο της επιστροφής στον ψυχρό πόλεμο. Αυτά που είπατε πρώτα πάρουμε πολύ στα σοβαρά. Ο κύριος Γκάλερ ανέφερε αυτή την παλιά ιστορία τη ζώνη ελευθερών πορείου και ήμουν ένα από του ε, βουλευτέ που είχαν συμμετάσχει αυτή την προσπάθεια μαζί με Γερμανού συναδελφού από 25 χρόνια και τότε οι διοικούντε στην περιοχή ε, με μεγάλο ενθουσιασμό ασχολήθηκαν με αυτή την πρωτοβουλία. Έγινε και μια διεθνή διάσκεψη εκεί όμω. Ποτέ δεν ήρθε η άδεια και το πράσινο φω από την Μόσχα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που περισσότερο με ανησυχεί είναι το ότι δεν υπάρχει κάποιο είδου ισορροπία μεταξύ των στρατηγικών σχεδίων της Μόσχας και της αντίδρασης της Δύσης. Τόσα χρόνια βλέπουμε αυτόν τον εξυγχρονισμό, αυτή την στρατηγική, από τότε που ανέβηκε στην εξουσία ο Πούτιν. εντύπωσή μου είναι ότι αμελούμε. Και δεν τα παίρνουμε στα σοβαρά όλα αυτά. Γιατί το δίδαγμα που πρέπει να αποκρούσουμε από όλα αυτά είναι ότι ο στρατηγικός στόχος της ε, Ρωσίας είναι να υπονομεύσει την ε, αρχιτονική ασφάλεια του ΝΑΤΟ και να στήσει μια δική της αρχιτονική. Το δεκίνητρο του κυρίου Πούτιν, πέστε μου τη γνώμη σας όμως αυτό, δεν είναι, δεν είναι στρατιωτικό, αλλά μάλλον πολιτικό. Θέλει να γκρεμίσει την αξιοπιστία που υπάρχει για τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Βαλτικής, ότι δηλαδή δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να υπερασπίσει τα πιο μακρινά του μέλη, τα πιο ευάλωτα. Θέλει επομένως να ταπεινώσει και να αποκυρώσει ούτως ή διεθνώς το να το Και γι' αυτό και δημιουργεί αυτή την καινούργια ζωή την παράθεση στην περιοχή και αναφέρει την αστάθεια. Και αποσταθεροποίηση όμω είναι πολύ ενισχυτικά όλα αυτά τα στοιχεία για το πόσο αποτελεσματικά μπορούν να καλύψουν την περιοχή της βαλτικής και ρωσικής δυνάμεις. Και άρα αναδείτε το πρακτικό ερώτημα. Αν υπάρξει κάποιο είδου επίθεση το ΝΑΤΟ χρειάζεται ταχεία ανάπτυξη επιπλέον δυνάμεων και εξοπλισμού υλικού. Πώς θα γίνει αυτό στη Βαλτική, αφού καλύπτεται τόσο καλή Βαλτική από τους Ρώσου, Είναι επομένω το δίλημα το εξή. Να φέρουν εκεί ένοπλες δυνάμεις ή του ΝΑΤΟ εκεί που χρειάζονται ή φοβόμαστε το ότι θα προκύψει προστριβή και σύγκρουση με τις ρωσικές δυνάμεις. Επίσης, σε σχέση με τον υβριδικό πόλεμο. Σας ευχαριστώ που το αναφέρατε. Ακριβώς, η ουσία αυτής της τακτικής είναι η αμφισημία, η αμφιβολία. Το να σπείρει κανείς εσωτερικές προστριβές, έτσι θα ξεκινήσει εκεί. Μετά πάμε στην αιματοχυσία και κατόπιν για να ειρηνεύσουν δήθεν την ε, περιοχή θα εισβάλλουν οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανεί μια πλήρη απάντηση. Εσείς τι λέτε. Η γραμματεία δεν είναι βέβαιο. Κύριε Μαζουράνη, ζητήσατε το λόγο. Αν ναι, τον έχετε. Thank you very much. Όχι, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω να μιλήσω. Σας ευχαριστώ, λέει ο βουλευτής. So I would like to, to also to, to put my... Και εγώ έχω ένα ερώτημα προς τον κύριο Μπερνιέ. Όσον αφορά την ανάπτυξη όπλων από πλευρά τη Ρωσία για το οποίο μας μιλήσατε ακόμα και αν αυτή η ανάπτυξη λαμβάνει χώρα σε ρωσική επικράτεια θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αυτό γιατί θα πρέπει να παρακολουθήσουμε το πώς εξελίσσονται τα πράγματα πώς αναβαθμίζεται εκεί ο εξοπλισμός. Πάντως, εμείς έχουμε σκεφτεί τα πιθανά σενάρια εκεί που είναι ούτως πίν περιοχές που έχει που εκκρεμεί κάποια σύγκρουση αυτό που λέγεται frozen conflict. Ότι ως αιτία στην Αμχαζία, Δηλαδή το τι δημιουργούν οι Ρώσοι εκεί που δεν είναι επικράτεια του κράτους τους, εκεί όμως που θέλουν να έχουν κάποιο είδου ε, πολιτικά κέρδη και εκεί όπου υπάρχουν διαφορετικές εναλλακτικέ για το τι θα κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις. Εκεί δηλαδή που θα είναι ευπρόσδεκτες από τον πληθυσμό. Ακριβώς όπως έγινε και στην Ουκρανία. Με αυτήν την μακρά περίοδο προπαρασκευής. Και βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα τώρα στην ε, Μολδαβία και προβληματιζόμαστε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη συνολικά, σφαιρικά τη στρατηγική της Ρωσίας. Η στρατηγική πλευρά των πραγμάτων είναι μόνο μία πλευρά του σενάρια. και θα πρέπει να δούμε το ότι σε επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το 2005-2007 περιγράφεται αυτή η τακτική, δηλαδή το πώς θα ανακτήσουν την επιρροή τους σε περιοχές που ανήκαν στην Σοβιετική Ένωση. Σοβιετική Ένωση ή τέλος πάντων στο Σοβιετικό Μπλοκ. θα πρέπει επομένω και εμείς να αντιδράσουμε με ένα σύνθετο τρόπο σε αυτά τα σύνθετα σχέδια. Παρακαλώ λάβετε το λόγο να απαντήσετε με την ίδια σειρά που κάνετε τις εισηγήσεις και αν μπορείτε καλύψτε όλες τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις. Πρώτος ο κύριος Παχόλσκι. Ενδιαφέρουσες όλες οι ερωτήσεις. Να σας απαντήσουμε τις ερωτήσεις. Καταρχήν το κατά πόσο υπάρχουν ενδέξεις ή συμπτώματα που αφορούν την ενδεχόμενη ανάπτυξη ενός πυρηνικού πολέμου σε αυτή την περιοχή. Πιστεύω ότι γνωρίζετε ότι στο ΝΑΤΟ ε, γίνονται τέτοια θέματα, δεν τα συζητάμε τώρα, αλλά εγώ θα μιλήσω από μια άλλη οπτική γωνία. υποθετική περίπτωση ότι ένα τέτοιο βήμα θα γίνει από τη Ρωσική Ομοσπονδία μπορεί να διαιρεθεί ε, στο ενδεχόμενο να γίνει απροκάλυπτα ή να γίνει συγκαλυμμένα. Και ε, υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία αναμένουμε από τη Ρωσία και έχουμε κάποια σενάρια σχέση με την ε, δική μας ε, πιθανή αντίδραση. Το δεύτερο σχόλιο είναι από καθαρά επιχειρησιακή οπτική γωνία. Ε, σημαντικό είναι το γεγονός ότι μπορούν πράγματι να χρησιμοποιηθούν ε, τέτοιου είδους ε, όπλα, να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε αυτή την περιοχή. Υπάρχει πρόβλεψη για κάτι τέτοιο. Άρα, στο πλαίσιο αυτό γίνεται ένα τεράστιο θέμα που δυστυχώς δεν είναι ιδιαίτερος επίκαιρο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ε, ε συζήτησης. Δηλαδή το πόσο διαφανή είναι τα, πόσο διαφανές είναι το πλωστάσιο, το πυρηνικό πλωστάσιο της Ρωσίας προς τα έξω και υπάρχουν ισχυρισμοί ότι θα πρέπει το ΝΑΤΟ να κάνει κάτι, να κάνει κάποιο βήμα πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για το ζήτημα της διαφάνειας. Αλλά υπάρχουν μικρές πιθανότητες να αλλάξει αυτή η κατάσταση σε σύντομο χρόνο, αλλά με όρους ακριβώς διαφάνειας ε, ή με όρους περιορισμού των μείωση των κινδύνων σε σχέση με το πώς χειρίζεται ε, η Ρωσία το θέμα του πυρηνικού οπλοστασίου. Είναι κρίσιμη σημασία στο ζήτημα αυτό. Το τρίτο σημείο αφορά το εξής. στο, στην περίπτωση που ισχύσει αυτό το υποθετικό σενάριο ενό ε, πυρηνικού πολέμου υπάρχουν ε, υπάρχουν ε, πολλοί τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ρωσία τα όπλα αυτά στην περιοχή αυτή η ανάπτυξη ενός πυρηνικού οπλοστασίου ενδεχομένω θα συνοδεύεται από μια από, από ένα σκεπτικό οικονομίας του πεδίου μάχης. Ε, θα πρέπει δηλαδή τα όπλα αυτά να επιφέρουν επιπρόσθετα ωφέλη για τη Ρωσία. Το θέμα είναι πώς ε, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα σύνορα με τη Ρωσία ε, από μια εθνική προοπτική καταβάλουμε κάθε τη προσπάθεια. Στο πλαίσιο του υβριδικού σεναρίου το ζητούμενο δεν είναι να υπάρξουν εθνικές λύσεις αλλά ολοκληρωμένα και στέρεα συστήματα αντίδρασης. Ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει κάποια βήματα. Αλλά από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ έχουν προκύψει κάποια άλλα επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στο επίπεδο μιας έγκαιρης προειδοποίησης ε, ή στο επίπεδο κάποιων ε, ενδείξεων βάσει των οποίων ε, θα μπορούσαμε να κινηθούμε, να αντιδράσουμε ή να προσλάβουμε τις προθέσεις της Ρωσίας. Αλλά εδώ μπορούν να γίνουν πολλές βελτιώσεις. especially uh, Έγγραφο της ε, Βιέννης ε, εφαρμόζεται μεν, αλλά όχι πλήρως ε, από τη Ρωσία. Όλες τις υποχρεώσεις λοιπόν δεν εκπληρούνται πλήρως και αυτή είναι μια επιπλέον πρόκληση που αφορά την αύξηση της διαφάνειας και την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή. Έγινε ένα σχόλιο προηγουμένως σε σχέση με το πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τη διευρυμένη παρουσία ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή. Ε, εγώ δεν θέλω να το υποτιμήσω, αλλά θα έπρεπε να το εξάσουμε από μια επιχειρησιακή οπτική. μιλώντας για αυτό το ευρυδικό μοντέλο, ε, υπό την έννοια της απόκτησης κάποιων ε, επιπλέον πλεονεκτημάτων στην περιοχή, ε, η παρουσία στο πεδίο της μάχης ε, στρατικών δυνάμεων στην Πολωνία και στη Βαλτική είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο σε όλους αυτούς τους υπολογισμού. Άρα, όπως είπα στην ομιλία μου, θα έπρεπε να ακολουθήσουμε ε, την, ε, να τηρήσουμε την αρχική μας απόφαση να αναπτύξουμε, να έχουμε μια ισχυρή παρουσία στην ανατολική μας πτέρυγα υπάρχουν κάποια τάγματα εκεί, υπάρχει, υπάρχει μια στρατιωτική παρουσία η οποία είναι αρκετά σημαντική. Όσον αφορά τα, την πυραυλική άμυνα, βεβαίως θα ήταν ιδεώδες να υπήρχε μια τέτοια προσέγγιση εκ μέρους του ΝΑΤΟ, δηλαδή μια αύξηση του των δυνατοτήτων άμυνας του ΝΑΤΟ. Ε, ε, το θέμα αυτό είναι, βεβαίω θα πρέπει να έχει μια πολιτική συνένεση εντό του ΝΑΤΟ. Πώς δηλαδή ε, σε ποιο επίπεδο θα εντερωθούν, θα αναπτυχθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Έχουμε κάποιες εμπειρίες τα περασμένα χρόνια όσον αφορά την περιοχή της Ανατολίας στην Τουρκία ε, και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στο επίπεδο της άμυνας ε, και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά το, τις δυνατότητές μας ε, την εναέρια, την αεροπορική άμυνα, όχι μόνο στην περιοχή αλλά γενικότερα αλλά προφανώς θα υπάρξει μια υποστήριξη από την Πολανία γιατί εμείς ε, θα επενδύσουμε πολλά σε αυτή την ε, προσπάθεια τα επόμενα χρόνια. Η Λιθουανία και οι άλλες βαλτικές χώρες επίσης προτίθενται να επενδύσουν εδώ στην αντιπυραυλική άμυνα και ε, το θέμα είναι πώς ε, μπορεί να γίνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει ληφθεί μια τέτοια απόφαση στις Βρυξέλλες, όχι ε, ίσως ίσως αυτή την αίθουσα, αλλά στο πλαίσιο άλλων θεσμικών οργάνων. Το τελευταίο ερώτημα ήταν τι μπορεί να γίνει στην περιοχή της ε, Βαλτικής. Εδώ υπάρχουν πολλές προκλήσεις από στρατιωτική άποψη. Ε, υπάρχουν ορισμένε απαντήσεις σε σχέση με το τι σημαίνει επίθεση και άμυνα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα ετοιμότητας των ε, δυνάμεων του ΝΑΤΟ που θα είναι η αρχική μας δύναμη για, εφόσον ισχύσουν τέτοιου είδους σενάρια, δηλαδή η δύναμη απόκρισης του ΝΑΤΟ και οι αποφάσεις που έγιναν στη Βαρσοβία, ε, αλλά που ελήφθησαν στη Βαρσοβία αλλά και μετά, ήταν προσανατολισμένες προς μια βελτίωση ακριβώς του χρόνου μετακίνησης των δυνάμεων αυτών προς την ε, περιοχή ε, εδώ βέβαια πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα σε εθνικό επίπεδο, όχι μόνο στην Πολωνία, αλλά και, στις ε, ε, και στη Λιθουανία και στις βαλτικές χώρες γίνονται προσπάθειες που περιλαμβάνουν και τις, τη βελτίωση των υποδομών, ούτω ώστε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα μια ταχεία απόκριση. Δεν πρόκειται όμως μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και άλλα στοιχεία που αφορούν την στρατηγική και όπου η ενίσχυση των δυνάμεων ε, θα είναι δυνατή όταν υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή ε, όσον αφορά το προγραμματισμό των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και βεβαίως ε, υπάρχουν κάποια σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν Ε, όσον αφορά την ενίσχυση της δικής μας θέσης, τόσο την πυρηνική, το πυρηνικό όσο και το συμβατικό πλωστάσιο, και γίνονται κάποιες σκέψεις πώς ε, μπορούν οι ενισχύσεις να φτάσουν στον κατάλληλο χρόνο και στον κατάλληλο τόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Να ζητήσω τώρα από τον κύριο Πετράητης να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ επίσης πολύ για τις δύσκολες, θα έλεγα, αυτές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω με τη σειρά που ετέθησαν. Και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, αν δεν απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Προσπάθησα να τις καταγράψω πάντως όλες. Από όσο κατάλαβα, η πρώτη είχε να κάνει με αυτό που ονομάσατε Green Polite Men, με τους στρατιώτες αυτούς. Είναι ένα από τα νέα δόγματα που χρησιμοποιούνται πλέον από τη Ρωσία. Ουσιαστικά, Πιστεύουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο οι Ρώσοι χρησιμοποιούν με φυΐα την εμπειρία του παρελθόντος. Πρόκειται ουσιαστικά για τη χρησιμοποίηση μισθοφόρων, τη χρησιμοποίηση στρατιωτών από ιδιωτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ακριβώς αυτό έγινε με την Ουκρανία και την Κρυμαία. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία προσπαθεί να δει αν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο και περισσότερο τους πόρους αυτούς και δεν γνωρίζουμε τελικά ακριβώς ποιος βρίσκεται πίσω από τις επιχειρήσεις αυτές γιατί καταλαβαίνετε ότι ε, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ε, κατ' επάγγελμα κάνουν ε, τη δουλειά αυτή, μπορεί να το διασκεδάζουν κιόλα, να το θέσω έτσι, και βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Η Ρωσία χρησιμοποιεί ένα τέτοιο νέο δόγμα και χρησιμοποιεί αυτές τις ιδιωτικέ υπηρεσίες τελικά τις στρατιωτικές με τρόπο ιδιαίτερα αποτελεσματικό, όσον αφορά τα νέα όπλα και πιο συγκεκριμένα το σύστημα βαλιστικό πυράβλων Ισκαντερ. Οι Ρώσοι ήδη έχουν κάνει πριν από 3-4 χρόνια κάποιες ανοιχτές δηλώσεις. Λέγανε ότι επρόκειτο να χρησιμοποιήσουν σε όλες τις ταξιαρχίες τους και μέχρι το 2018 συστήματα Ισκαντερ. Αν δούμε λοιπόν την ταξιαρχία αυτή που έχουν στο Καλίνιγκραντ, αυτή μπορεί ενδεχομένως να μην έχει ακόμα εξοπλιστεί αναλόγως, αλλά πρόκειται να συμβεί. Αυτό θα είναι αποτελεμιστικό του χρόνου ή μετά από κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα θα δούμε και εκεί τη χρησιμοποίηση συστημάτων Ισκαντερ. Όσον αφορά την δυνατότητα μεταφοράς και παράδοσης πυρηνικών κεφαλών στην περιοχή, και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Τα περισσότερα οπλικά συστήματα της Ρωσίας προέρχονται από τη Σοβιετική εποχή και οι ε, Ρώσοι ακόμα εμπνέονται τελικά από την εποχή αυτή όπου ε, όλα τα οπλικά του συστήματα τα παρήγαγαν με δύο αν θέλετε εκδοχές. Υπήρχε πάντα και η πυρηνική εκδοχή. Αν μιλούμε για παράδειγμα για τα βαλιστικά συστήματα 300, M300, τότε αυτά ή τα S300, με συγχωρείτε, ή τα S400 θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην είναι μόνο συμβατικά όπλα, αλλά να μπορούν να μεταφέρουν και πυρηνικέ κεφαλές. Συνεχίζουν λοιπόν οι Ρώσοι και βασίζονται σε μια προσέγγιση που είχαν από την περιοχή της Σοβιετικής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα την μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων. Η Λιθουανία είναι μια χώρα που χωρίζει βασικά την υπηρετική Ρωσία από το Καλίνιγκραντ. Υπάρχουν προφανώ συγκεκριμένε συμφωνίε μεταφορά και μετακινήσεων μεταξύ Λιθουανία και Ρωσία που βασίζονται σε μια συμφωνία που υπεγράφει πριν από μερικά χρόνια όταν η Ρωσία άρχισε να αποσύρει δυνάμει από τη Γερμανία. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι κανόνες στρατιωτικών μεταφορών, στρατιωτικών κινήσεων, οι οποίοι ε, κανόνες λειτουργούν καλά, αλλά που τελικά από ό,τι φαίνεται δεν χρησιμοποιούνται από τους Ρώσους. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια είναι ότι όλες οι παραδόσεις, οι μεταφορές που έχουν γίνει από τους Ρώσους είχαν να κάνουν κυρίως με μη στρατιωτικό υλικό με εξοπλισμούς που θέλουν να εγκαταστήσουν οι Ρώσοι στο Καλίνιγκρατ, αλλά που δεν είχαν κάποια στρατιωτική χρήση. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι οι Ρώσοι εφόσον θέλαν να εγκαταστήσουν στο Καλίνιγκραντ στρατιωτικό εξοπλισμό θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη θαλάσσια οδό. Και αυτό άλλωστε έχουν κάνει οι Ρώσοι με τα συστήματα Ισκαντερ και σε άλλες περιοχές όπου τα έχουν εγκαταστήσει. Υφίστανται λοιπόν οι κανόνες αυτοί, δεν τίθενται να αμφιβόλω από καμία πλευρά. Εμείς θεωρούμε πάντως ότι οι στρατιωτικές αυτές μεταφορές μπορούν να αποτελέσουν απειλή για τη Λιθουανία. Όσον αφορά πάντως τη μεταφορά όπλων ή ευαίσθητων, αν θέλετε, αγαθών, φαντάζομαι ότι η Ρωσία δεν θα προτιμήσει την οδική οδό, τη χερσαία οδό, αλλά θα προτιμήσει την ενέργεια οδό και τη θαλάσσια οδό. Τώρα, Όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων, προφανώς υπάρχουν και εκεί συμφωνίες με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Συγκεκριμένες συμφωνίες όσον αφορά την υιοθέτηση των συνόρων. Εγώ σε μερικές εβδομάδες θα πρέπει να πάω στη Μόσχα γιατί είμαι μέλος της Λιθουανικής Αντιπροσωπείας για την διαπραγμάτευση της διαδικασίας αυτής. Προσπαθούμε τη διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί του χρόνου. Αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα, έχουμε κάποιες διαφωνίες αλλά θεωρούμε ότι πολύ σύντομα θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία αυτή και θα έχουμε ένα σωστά όριοθετημένο χερσαίο σύνορο με την ε, Ρωσία. Όσον αφορά την ε, στρατιωτική λεγόμενη διαφάνεια, το ανέφεραν και αυτό οι συναδελφοί μου. Δυστυχώ πρέπει να αποδεχθούμε το ότι η Ρωσία κάνει πάρα πολλά πράγματα προκειμένου να καταστρέψει, αν θέλετε, το εφιστάμενο στρατιωτικό καθεστώς στην Ευρώπη. Θυμάστε το είχε πει αυτό και ο πρόεδρος Μετβέντεφ στο παρελθόν. Είχε πει ότι η Ρωσία δεν ήταν ικανοποιημένη με το εφιστάμενο ευρωπαϊκό στρατιωτικό καθεστώς και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσει η Ρωσία, να θετήσει, αν θέλετε, το έγγραφο της Βιέννη, προκειμένου να ταχθεί κατά του ευρωπαϊκού στρατιωτικού καθεστώτος. Βλέπουμε ότι οι Ρώσοι θέλουν να επικαιροποιήσουν το έγγραφο αυτό, τώρα εν 2016 όσον αφορά τη στρατοτική διαφάνεια σε διμερέστορο επίπεδο. Βασιζόμενοι στο έγγραφο της Βιέννης έχουμε διμερεί στρατιωτικές συμφωνίες με τη Ρωσική Ομοσπονδία για την ανταλλαγή στρατιωτικών μονάδων παρατηρήσεων και επιθεωρήσεων. Μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο δικές τους μονάδες να έρθουν σε εμά και το αντίστροφο. Και μπορούμε και εμείς κατά αυτόν τον τρόπο να πηγαίνουμε στο Καλίνιγκρατ. Δυστυχώς το 2011, αν δεν κάνω λάθος, οι Ρώσοι με δική του πρωτοβουλία ακύρωσαν την υφιστάμενη αυτή διμερή συμφωνία και επί του παρόντος δεν έχουμε κανένα διμερές σύμφωνο που να μας επιτρέπει τέτοιες ανταλλαγές. Οι Ρώσοι από ό,τι βλέπετε κάνουν κάθε τι το δυνατό προκειμένου να ενισχύσουν την παρουσία του στη Βαλτική και θέλουν αυτή να γίνει πραγματικότητα. Αν λοιπόν οποιαδήποτε χώρα τελικά αποφασίσει ότι ε, χρειάζεται μια επιπλέον δική μας στρατιωτική παρουσία στην περιοχή κοντά στο Καλίνιγκρατ εξαιτίας της Ρωσίας, τότε αυτή θα πρέπει να εισακουστεί. Έχουν, πει, έχουν κάνει διάφορες ψευδείς δηλώσεις οι Ρώσοι. Εγώ θα έλεγα ότι στη Λιθουανία έχουμε δημιουργήσει πολλές επιπλέον ταξιαρχίες και στρατιωτικές μονάδες. Ο Υπουργός μας και η κυβέρνησή μας έχει εγκρίνει την δημιουργία των νέων αυτών μονάδων και έχει γίνει μια μεταφορά των μονάδων αυτών στα σύνορα με το Καλίνιγκραντ. Δεν αληθεύει λοιπόν αυτό το οποίο ακούστηκε πριν από λίγο ότι δεν έχουμε μια κάποια στρατηγική δραστηριότητα, στρατιωτική με δραστηριότητα στη Λιθουανία. Προφανώς επενδύουμε στην αμυντική μας βιομηχανία και επενδύουμε σε εγκατάσταση στρατιωτικών μονάδων. Όσον αφορά τώρα το ότι ε, οι ρωσικές στρατιωτικές μονάδες διακατέχονται από όλο και μεγαλύτερο επίπεδο επαγγελματισμού. Αυτό αληθεύει. Ο Υπουργός Άμυνα της χώρας με ιδιαίτερη περηφάνεια δήλωσε ότι ο αριθμός των επαγγελματικών οπλητών έχει ξεπεράσει πλέον τους στρατευμένου νέους της χώρας και ότι υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες μονάδες, ιδίως της ταχείας εξάπλωσης και αντίδρασης, που απαρτίζονται πλέον σχεδόν αποκλειστικά από επαγγελματίε οπλίτες, από επαγγελματίε στρατιώτες. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σε πανρωσικό επίπεδο έχουν ξεκινήσει μια πολύ ε, αποτελεσματική εκστρατεία πρόσληψης νέων ε, στρατιωτών. Και κατά αυτόν τον τρόπο βλέπετε ότι εκμεταλλεύονται όλες τις ε, δυνατότητες που τους δίνονται με τη χρησιμοποίηση όλο και περισσότερων νέων ε, επαγγελματιών στρατιωτών. Όσον αφορά τώρα την τοποθέτηση μονάδων πυράβλων Patriot στη δική μας την περιοχή, θα ήμουν ευτυχή να συνέβαινε κάτι τέτοιο, αλλά πάλι αυτό εξαρτάται από τι αποφάσει που θα πρέπει να λάβουμε, που θα βασίζονται σε συγκεκριμένε εκτιμήσει πώς θα καταφέρουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε τα νέα όπλα που έχουν οι Ρώσοι, πώς θα καταφέρουμε να σπάσουμε το δόγμα α2AD των Ρώσων, αυτό το νέο δόγμα περιορισμού, η επαγόρευση της πρόσβασης. Και καταλαβαίνετε ότι ε, το δόγμα αυτό το εφαρμόζουν οι Ρώσοι όχι μόνο στην περιοχή της Βαλτικής, αλλά ακόμα και στην ε, περιοχή της Ασίας. Θα μπορούσαμε πάντως να αντιμετωπίσουμε τη δική τους ε, γεωγραφική κάλυψη, τη δική τους ε, ασπίδα με μια δική μας αντιπυραυλική ασπίδα. Αυτό εξαρτάται πάντως από τη δική μας την ε, στρατιωτική εμπειρογνωμοσύνη, τι όπλα θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, πόσο γρήγορα θα καταφέρουμε να αναπτύξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα αυτά. Εξαρτάται λοιπόν πάλι αυτό από τις στρατιωτικές συμβουλές που θα πρέπει να μας δώσει το ΝΑΤΟ. Όσον αφορά τώρα τι τελευταίε ερωτήσει που ακούσαμε, ενδεχομένω να μην καταφέρω να απαντήσω κάποιες από αυτές, γιατί ουσιαστικά απευθύνονται περισσότερο στον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ, τα όσα είπατε για τον Ιβρετικό πόλεμο κτλ. Ωστόσο, θεωρώ ότι γίνανε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσε παρατηρήσεις για τη ρωσική στρατηγική υποκατάσταση της παρουσίας τη Αμερική στην Ευρώπη θα ήθελα να αναφερθώ σε μία εκδήλωση στην οποία είχα πάει πριν από 4 ή 5 χρόνια, όταν τότε ακόμα υπήρχε μια κάποια συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας και είχαν γίνει τότε κάποιες συζητήσεις για δόγματα στρατιωτικά με στρατιωτικούς από τη Ρωσία που είχαν έρθει σε αυτή την εκδήλωση. Και δόθηκε μια δεξίωση το βράδυ της συνεδρίασης αυτής και ξέρετε ότι πολύ συχνά διεξάγει κανείς μια συζήτηση λίγο πιο χαλαρή κατά τη διάρκεια των κοκτέιλ αυτών των δεξιώσεων. Είπα λοιπόν τότε, είπε μάλλον ένας Ρώσος ότι το ΝΑΤΟ έχει ως στόχο τελικά να αποτρέψει τους Ρώσους και να καταφέρει να κρατήσει σε υποδέστερη θέση, αν θέλετε, τους Γερμανούς. Και αυτό υπόθηκε λοιπόν ανεπίσημα κατά τη διάρκεια της δεξίωσης αυτής, αλλά άμα το σκεφτείτε, ενδεχομένως θα μπορούσε όντως η Ρωσία να εξετάσει περισσότερο τη δυνατότητα μιας κάποιας ανεπίσημης ε, συμμετοχής στο ΝΑΤΟ. Κύριος Μπαρνιά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ για όλες σας τις ε, ερωτήσεις και το κοινό σημείο όλων να ρωτήσουν το τι θα κάνουμε για τόσα διφορούμενα σημεία, όπως δηλαδή τι γίνεται με αυτούς τους ιδιωτικούς στρατούς, τα πράσινα ανθρωπάκια και πώς θα μπορέσουμε κάπως να αντιδράσουμε. Τι θα γίνει με το ότι χρειάζεται ταχεία λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο από πλευρά του ΝΑΤΟ για τους πύραυλους ε, Ισκαντέρ και γενικότερα για τις ε, δυνατότητες των Ρώσων με τις ε, συμβατικές και τις ποινικές κεφαλές. Αυτά όλα γίνονται για στρατηγικού στόχου, αλλά επίση και για να ενισχύσουν αυτήν την ε, ατμόσφαιρα αμφιβολίας. Αυτό διαπνέει όλε αυτέ τι ενέργειε και αυτή είναι μια δυσκολία για μας γιατί εμεί δεν έχουμε τι πληροφορίε, ούτω ώστε γι' αυτό βρισκόμαστε σε κατάσταση αμφιβολίας. Επίσης το βασικό για μας και από πλευράς στρατηγικής και πολιτικοστρατηγικής είναι η ανθεκτικότητα του στρατού μας, της κοινωνίας μας, των πολιτικών οργάνων μας όσον αφορά τις πιθανότητες επίθεσης, όσον αφορά αυτή την ατμόσφαιρα αμφιβολίας, όσον αφορά τις υβριδικές δραστηριότητες. Όσον αφορά την σύγκριση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ με τις ρωσικές δυνάμεις στην Βαλτική. Όχι, για μας δεν έχει σημασία το να εξισώσουμε τις δυνάμεις μας με εκείνους όσους ταξιαρχείς και να παρατάσουν ή να αντιδρούμε μία σου και μία μου που λέμε, ε, ούτε να δαπανούμε όσο και εκείνη. Εμείς θέλουμε να τρίσουμε βήμα στην τακτική του, να διαλύσουμε πάσα αμφιβολία, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Θέλουμε να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα που στέλνουμε, θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά την κοινή γνώμη μας ε, και να έχουμε επομένω ε, γι' αυτό το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, αυτό το tripwire. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι στέρεο, στεγανό σύστημα. Και βεβαίω ε, όλα αυτά στηρίζονται και ώστε να έχουμε ε, καλές σχέσεις μεταξύ μας και με την κάθε φορά φιλοξενούσα εμάς χώρα. Τώρα, αναφέρθηκε το θέμα της συμβολικής χειρονομίας. Να ισχύει αυτό. Πολιτικά, στρατηγικά, πάρα πολύ σημαντικό και συμβολικά και στρατιωτικά, γιατί είναι θέμα αξιοπιστίας του συστήματος προειδοποίησης, του Tripwire. Θα πρέπει βέβαια όλα αυτά να είναι στρατιωτικά βιώσιμα. Εκεί δίνουμε το βάρος για το Tripwire. Τώρα όσον αφορά την πυραυλική άμυνα. Η άμυνα μας δεν στρέφεται κατά τη Ρωσία. Αυτό το έχουμε πει από τότε που ελήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. και το έχουμε παραλάβει. Παρά τα όσα λένε συνεχώς οι Ρώσοι. Πρώτα-πρώτα, δεν έχουμε στο ίδιο επίπεδο στρατηγικές ε, βλέψεις. Πάντως, όπως ξέρετε, στη φυσική Η κάθε δράση είναι η αντίδραση. Εμεί αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε αποτρεπτικό δόγμα. Για όλου αυτού του λόγου δεν ισχύει το ότι εμεί κάνουμε παιδιά και αυτό αποφάσισε και το, ΤΟΝΑΤΟ Να μην έχουμε πολλαπλασιασμό των πυράβλων και συγκεκριμένα όσον αφορά την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων που θα αναπτύσσαμε σε περίπτωση σύγκρουση δυσκολία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τις ρωσικές δυνάμεις και το διπλό ρόλο, τη διπλή φύση ε, των, οπλισμών του, δηλαδή συμβολικά και δεν συγγνώμη, συμβατικέ όπλα και πυρηνικά όπλα, αυτό μας απασχολεί. Μας αναφέρατε επίσης για τον εκφοβισμό και την ταπείνωση. Είναι σωστό ότι αυτά τα μετέρχονται. Αυτή είναι δύσκολη και για μας. Έχουμε αυτό το σενάριο της αναμέτρησης δυνάμεων, τον εκφοβισμό και την ταπείνωση. Οπότε έχουμε επιστρατεύσει ένα συγκεκριμένο οπλοστάσιο καθώς επίσης και την δύναμη ταχείας αντίδρασης όπως συζητήθηκε στην συνάντηση κορυφής και συνοδεύεται από τις δυνάμεις που ακολουθούν ταχεία αντίδραση. Έχουμε τα σωστά στάνταρ, σωστή ε, εκπαίδευση, την διαλειτουργικότητα ε, με τους εταίρους μας και μεταξύ μας τα κράτη-μέλη. Και πάνω σε αυτό ενεργούμε. Αυτό ως βάση. Έχουμε τώρα κάποιες άλλες ε, πιο τεχνικές ερωτήσεις και παρεμπιπτόντως πρέπει να σας πω ότι μετά το σχέδιο δράσης και της κορυφής είναι πάρα πολύ σημαντική η επιμελητία για όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Είναι πολύ σημαντική για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. για τις προμήθειες, για τα πυρομαχικά, για όλα αυτά, για τα καύσιμα. Και πώς συγκρατήσαμε τη δική τους δυνατότητα στον ίδιο τομέα. Αυτό καταλαβαίνω. Τι γίνεται στους λιμένες και λοιπά τι γίνεται όσον αφορά τη νομοθεσία για μεταφορά τοξικών υλικών, τι γίνεται με τη μεταφορά πυρομαχικών. Αυτά μας προβλημάτισαν βαθιά και έχουμε εμπειρογνωμοσύνη, γιατί έχουμε κάνει μια διαδρομή πολλών ετών. Και μας απασχολεί το θέμα και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε εθνικό επίπεδο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. αν φοβόμαστε τη σύγκρουση. Ήταν μια άλλη ερώτηση πολύ εύστοχη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε τη σύγκρουση. Για μας η αποτροπή, η πυρηνική αποτροπή ακριβώς αποσκοπεί στο να μην υπάρξει σύγκρουση. Να μην θεωρήσει ότι μπορεί να τα καταφέρει να, να ε, μας εκφοβήσει κάποιος ε, αντίπαλος. Εδώ και δύο χρόνια ασχοληθήκαμε με τον ε, υβριδικό πόλεμο. Εξού και η έννοια της ανθεκτικότητας που μας απασχόλησε η σχέση ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε εργαλεία και μέσα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα από πλευρά ε, άμυνα και ασφάλεια των κρατών μελών και των σύμμαχων. Έχουμε κάποιου ε, δείκτε, προειδοποιήσει για να μπορέσουμε να δούμε το πότε κάτι θα ξεκινήσει, το πότε κάτι θα συμβεί. Το βασικό στοιχείο, κύριε Πρόεδρε, είναι το ότι δεν βλέπουμε καμία αφαίρετη σχέση με την Ρωσία. το βασικό είναι να υπάρχει προβλεψιμότητα, όπως ισχύει σήμερα. Άρα, εμείς έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την άμυνά μας, για την προστασία των συμμάχων μας. Όμως, θα πρέπει να δούμε και το πώς θα βελτιωθεί και η πολιτική ατμόσφαιρα κάποια στιγμή στο μέλλον. Οπότε το τότε να δούμε πώ θα υπάρξει έλεγχο εξοπλισμών, ε, πώ θα συζητηθεί η υπόθεση τη εθνική κυριαρχία και τη διαφάνεια. Αυτά για το μέλλον. Η ε, Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε. Όλου ευχαριστώ που ήρθατε εδώ και κάνατε αυτέ τι ε, εισηγήσει. Σα ευχαριστώ και του συναδέλφου για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα όποτε χρειαστεί. Όποτε χρειάζεται θα το ξανασυζητούμε. Πάντως τώρα έχουμε ολοκληρώσει αυτό το θέμα στην ημερησία διάταξη και το επόμενο σημείο είναι ο διοικητής του στοιχειωτικού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε.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 Ladies Κυρίες και κύριοι, επιτρέψατε μου να καλωσορίσω τον ε, κύριο αντιστράτηγο, κύριο Αποκάνεν, έσ Πουκάνεν, που θα παρουσιάσει τον ε, ρόλο του στρατιωτικού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, θα ήθελα να σας καλησπερίσω όλους. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά για μένα που απευθύνομαι σε αυτή την Επιτροπή εδώ. Είναι μια ενδιαφέρουσα μέρα, όπως όλοι επιστώσαμε όταν ξυπνήσαμε. Και εγώ πολύ συχνά ανοίγω τις παρουσιάσεις μου λέγοντας ότι η κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη είναι σε, βρίσκεται σε μια ραγδαία αλλαγή. Ε, αλλά όπως και το πολιτικό κλίμα αλλάζει ραγδαία και πραγματικά δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, τι βρίσκεται στον ορίζοντα. Αλλά και τα θέματα ασφάλειας είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ε, ναι, μεν φοράω στρατιωτική στολή, αλλά θα μιλήσω για την ε, ήπια ε, πτυχή ε, του θέματος, σε αντίστοιξη με τους συναδέλφους. Έρχομαι πρώτη, ήρθα πρώτη φορά το 2000 στις Βρυξέλλες και ήμουν από τους πρώτους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που κλέθησαν να παρουσιάσουν τη στρατιωτική διάσταση. Τότε ε, είχαμε μία μόνιμη κατοικία ε, και ε, μπορούσα να πάω ε, με, να χρησιμοποιήσω ποδήλατο για να πάω στη δουλειά μου ε, και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ασφάλειας. Σήμερα έχουν αλλάξει όλα ριζικά. Ε, Βεβαίω, όλα αυτά τα σύνθετα μέτρα ασφαλείας είναι με δυσάρεστα αλλά αυξάνουν το βαθμό ασφάλειας. είναι ενδιαφέρον ε, βεβαίως να εργάζεται κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ορισμένοι λένε τι γυρεύουν οι στρατιωτικοί στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη αποσκοπεί στην ειρήνη. Αυτή είναι φυσική αντίθεση ορισμένων συναδέλφων. Αλλά μετά από μερικούς ε, μήνες υπήρξαν και κάποιες ε, γυναίκες που αποτάνθηκαν σε μας ε, και μας είπαν ότι είναι καλό που βρίσκεστε εσείς εδώ. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι εδώ στις ε, Βρυξέλλες και πραγματικά είμαι περήφανος που επελέγει εδώ εκ μέρους του στρατιωτικού προσωπικού. Ε, θα μείνω μέχρι το Μάη εδώ ως Διευθυντής του Στρατιωτικού Προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πολλά πράγματα ε, συνέβησαν από τότε που ξεκίνησα Βεβαίως, ε, ε, υπήρξαν πολλές σημαντικές εξελίξεις στο Brexit και οι εκλογές ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ζητήματα που θα έχουν, αν όχι άμεσες, τουλάχιστον έμεσες επιπτώσεις και στη δική μας δουλειά. Πολλά από τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι τώρα στο δικό μου επιτελείο που αποτελείται από 200 ε, πολίτες και στρατιωτικούς, πολιτικούς υπαλλήλου και στρατιωτικούς, αφορούν με την εφαρμογή της ε, συνολικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Εγώ έθεσα κάποιες προτεραιότητες ήδη από τον πρώτο χρόνο και μία από αυτές αναφέρθηκε ήδη η σφαιρά της παγκόσμιας στρατηγικής και το ζήτημα της εφαρμογής καθώς και η εξασφάλιση του ρόλου του, των στρατιωτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστήριξη δηλαδή στις διάφορες αποστολές ε, και επιχειρήσεις εκεί όπου ε, γίνονται, κυρίως σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως στην Αφρική. Μία παγκόσμια στρατηγική η οποία δημιουργήθηκε ε, από την ε, από τα Now, since, uh, running... την είπατε εκπρόσωπο ε, και εμεί εισφέραμε σε αυτήν και υποβάλαμε κάποιες ε, προτάσεις για θέματα στρατηγικής και για θέματα εφαρμογής της στρατηγικής αυτής και ήταν μια χαρά για μας να μπορούμε να παράσχουμε και τις δικές μας ε, ιδέες όσον αφορά το πρόγραμμα εφαρμογής ε, το οποίο συζητήθηκε σε πάρα πολλές επιτροπές ε, στο Συμβούλιο και είναι βεβαίως ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τα οποία λαμβάνονται υπόψη από όλες τις χώρες ε, μέλη και θα τεθούν και πάλι τα θέματα στην ε, προσεχή σύνοδο. Υπάρχουν έμεσες βεβαίως επιπτώσεις για το στρατιωτικό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως ε, διαβάσετε ήδη τη στρατηγική αυτή και έχετε γνώση της συζήτηση η οποία ακολούθησε όχι μόνο εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά και στις διάφορες ε, πρωτεύουσε των χωρών μελών. Και θα έλεγα ότι κάποιες επιπτώσεις που είναι πολύ προφανείς για μας σχετίζονται από τη μία με τις στρατιωτικές δυνατότητες όπου βεβαίως το στρατιωτικό προσωπικό εδώ παίζει έναν διδραματίζει σημαντικό ρόλο προσπαθώντας να ορίσει τις προϋποθέσεις των στρατιωτικών δυνατοτήτων που θα πρέπει να αναπτυχθούν. Και ε, στο επίπεδο των διαφόρων οργάνων ε, και της Επιτροπής ε, βεβαίως υπάρχει, υπάρχει μια συμμετοχή και των άλλων θεσμικών οργάνων αλλά και εμείς από τη δική μας πλευρά προσπαθούμε να ορίσουμε αυτές τις προϋποθέσεις ε, προσπαθώντας να αναλύσουμε διάφορα σενάρια καταρχήν και στη συνέχεια να διατυπώσουμε τις προϋποθέσεις και τις βασικές ε, παραδοχές ε, για τη στρατηγική μας και σε σχέση με τι θα κάνουμε τους προσεχείς μήνες και τα προσεχή έτη. Δεν είναι εξαιρετικά χρονοβόρο αυτή η διαδικασία, παρόλα αυτά χρειάζεται κάποιο χρόνο για να γίνει και ίσως κάποιος ε, σχηματίζει ε, ε, και, και εδώ το Υπουργείο Άμυνας παίζει έναν σημαντικό ρόλο και υπάρχει και ένας συντονισμός με τον ΝΑΤΟ γιατί στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιες ε, δυνατότητες που σχετίζονται με τις χώρες μέλη. Υπάρχει ένα, μια ενδιαφέρουσα πτυχή του θέματος της εφαρμογής που σχετίζεται με τις ε, δομές και υπάρχουν πολλές προσδοκίες ε, εν σχέση με την βελτίωση της, ε, το, της ε, πολιτικής και στρατιωτικής ε, συνέργειας μιας μεικτής συμμετοχής δηλαδή στις επιχειρήσεις του πολιτικού και του στρατιωτικού μέρους και του τρόπου με τον οποίο διεξάγονται. Θα έλεγα ότι η βασική παραδοχή για τον σχεδιασμό μας, για τον, για τον σχεδιασμό μας είναι ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια αποτελέσματα από τη μία είναι μέσα αποτελεσματική, από την άλλη δεν είναι εύκολο να υπάρξουν πόροι ε, εκ μέρου των χωρών μελών. Ε, θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι απτόρατο και να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ε, προσπαθούμε να δημιουργηθούν καλύτερες ε, συνέργειες μεταξύ ε, στρατιωτικών και του στρατιωτικού και μη στρατιωτικού μέρους στο επίπεδο των διαφόρων διευθύνσεων της Επιτροπής και ταυτόχρονα προσπαθούμε να παράσουμε καλύτερη υποστήριξη στις επιχειρήσεις και τις αποστολές μας. Και το πρώτο μου έβριμα, το οποίο βασίζεται στην ε, παρουσία μου εδώ των πέντε μηνών, είναι ότι υπάρχει μια σοβαρή πρόκληση εν σχέση με την σχέση, μεταξύ ε, ε, Βρυξελών και, και αποστολών εκπαίδευσης ε, στις ε, ε, διάφορες χώρες, στη Σομαλία, την Αφρική κλπ. υπάρχει από τη μία πλευρά άσκηση πολιτικού ελέγχου και αυτό δείχνει σε μια κατάσταση όπου η στρατιωτική επικεφαλής καλούνται να πάρουν μια απόφαση, αλλά τελικά δεν γνωρίζουν σε ποιον αποτανθούν, γιατί κανείς δεν είναι υπεύθυνος. Υπάρχει λοιπόν, ε, λείπει εδώ ένας συνδετικός ε, κρίκος, υπάρχει λυπής υποστήριξη ε, εδώ και αυτό είναι το πρώτο θέμα το οποίο θα έπρεπε να δούμε, δηλαδή να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα για το στρατιωτικό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να αναλάβει το συντονισμό με τις Βρυξέλλες. Αυτό σημαίνει ότι τα διάφορα ε, στρατιωτικά επιτελεία ε, ε, συχνά δεν θα πρέπει να κάνουν το συντονισμό μεταξύ Αφρικής και Βρυξελών, αλλά, θα πρέπει να, αλλά αυτό θα γίνεται μέσω ενός άλλου και θα υπάρξει και συνεχής παροχή υποστήριξη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, το πρώτο θέμα το οποίο θα πρέπει ακριβώς να ορίσουμε. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με τις ε, παρούσεις μας ε, δυνατότητες, ε, εφόσον αποκτήσουμε αυτή την αρμοδιότητα. Τώρα, όσον αφορά τη συνέργεια μεταξύ μη στρατιωτικού και στρατιωτικού βραχίωνα, έχω καμιά φορά την εντύπωση ότι ε, δεν καταλαβαίνει κανείς ε, περί τίνος ομιλούμε. Ε, το μη στρατιωτικό, civilian, είναι ένας όρος που συχνά παρανοείται. Εμείς έχουμε μια τέτοια μορφή συνεργασίας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά μη, μη στρατιωτικά όργανα. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε κάνουμε με τους όρους της παροχής στρατιωτικής ε, δυνατότητας συμπεριλαμβάνει ακριβώς και αυτό τον, ε, τη μη στρατιωτική ε, πτυχή. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο λειτουργεί καλά είναι η συνεργασία εντός της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Έχουμε το κέντρο παροχής πληροφοριών που αποτελείται από εμπειρογνώμονες, από τις ε, εμπειρογνώμονες από διάφορες υπηρεσίες ε, πληροφοριών. Και έχουμε επίσης ένα ε, διευθυντήριο στρατιωτικής υπηρεσίας παροχής συγκέντρωσης πληροφοριών. και το προϊόν από τις δύο αυτές υπηρεσίες, δική και μη στρατιωτική από τις δύο αυτές υπηρεσίες πληροφοριών, ε, χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο. Και ίσως ε, πραγματικά είναι μοναδικό αυτό ε, στον κόσμο και οδηγεί σε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχουμε όλο και μεγαλύτερη ζήτηση και όλο και αιτήματα, μάλλον έχουμε όλο και περισσότερα ετήματα, συγγνώμη, να ασχοληθούμε και να έρθουμε σε έναν διάλογο με την Επιτροπή εν σχέση με τον εξοπλισμό, όχι τον καθαρά στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά για παράδειγμα την υποστήριξη του καθημερινού βίου, την, ε, ε, τις στολές κλπ. Επίσης υπάρχουν κάποια τμήματα κατάρτισης που έχουν ανάγκη όλο αυτό το υλικό. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν οι τρόποι να... Υπάρχουν κάποιες ε, οικονομικές διευθετήσεις και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία δεν μπορούν εύκολα να επιληθούν μέσω των υφιστάμενων δομών αλλά εάν υπάρχει παρκής πολιτική βούληση μπορούν ε, να αξιοποιηθούν οι δομές για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών αποστολών. Γιατί ναι, μεν εκπαιδεύουμε ε, στρατεύματα, αλλά την... Ε, Δεν έχουμε πάντα τη δυνατότητα να έχουμε τα τέλεια αποτελέσματα. Από δομικής τώρα πλευράς, αν θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε τις συνέργειες αυτές, θα πρέπει να λάβουμε πιο συγκεκριμένο ρόλο όσον αφορά τον κλάδο του ελέγχου. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε κάποιες πιο μόνιμες δομές εδώ στις Βρυξέλλες σε σχέση με τις αποστολές και τις επιχειρήσεις κατάρτισης. Αυτός από μόνος του είναι ένας στόχος. Αν δούμε τώρα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τις κινητικές αυτές επιχειρήσεις, την Άλθεα, για παράδειγμα, καθώς επίσης και τις επιχειρήσεις που διεξάγουμε μαζί με το ΝΑΤΟ ή την επιχείρηση Αταλάντα ή Σόφια, όπου την διοίκηση έχει η ουσιαστικά Ευρωπαϊκή Ένωση, βασιζόμαστε πάλι σε διευθετήσεις και κανονισμούς του ΝΑΤΟ. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες στρατιωτικές απαιτήσεις για βελτίωση της κατάστασης. Να έχουμε δηλαδή μια πιο μόνιμη δομή που θα μας επέτρεπε να διευκολύνουμε την πρώιμη, πρώτερη μάλλον προκαταρκτική σχεδίαση μιας αποστολής και μιας επιχείρησης. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρναμε να είχαμε μια πιο μόνιμη δομή εδώ πέρα στις Βρυξέλλες που θα μας επέτρεπε να σχεδιάζουμε καλύτερα και των προτέρων της επιχείρησης. Το ζήτημα όμως αυτό έχει μια έντονα πολιτική διάσταση. Εγώ παρουσιάζω μόνο, θέλετε, την δική μου στρατιωτική οπτική γωνία. Έχω εντοπίσει την ανάγκη αυτή, επιθυμούμε να υλοποιηθεί στο μέλλον εξαρτάται σαφώς από την πολιτική βούληση των κρατών μελών. Να δημιουργηθεί δηλαδή, το παραλαμβάνω, αυτή η μόνιμη δομή πέρα από το στρατιωτικό επιτελείο που έχουμε ήδη στις Βρυξέλλες και έχοντας κατά νου τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια του δικού μας του επιτελείου. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και περιορισμοί στις δικές μας αρμοδιότητες και όσον αφορά την, α, τους εξοπλισμούς ή τη στελέχωση των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να στελεχώνουμε καλύτερα και να εξοπλίζουμε καλύτερα τις επιχειρήσεις αυτές ήπια δύναμη, όπω λέγονται, που έχουν να κάνουν κυρίω με κατάρτιση. Θα δούμε τώρα πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώ θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τη στρατηγική αυτή και εμεί ε, προφανώ είμαστε εδώ πέρα για να υποστηρίξουμε του ε, πολιτικού προϊστάμενους μα. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα, Πρόεδρο. Σα ε, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Στάτιν έχει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Στρατηγέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα σήμερα. Είστε ύπατο εκπρόσωπο λοιπόν των στρατικών δυνάμεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχω να σα κάνω μια ερώτηση η οποία προκύπτει πολύ συχνά. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε, δεχόμαστε στην Επιτροπή μας ε, υψηλά ιστάμενους ε, αξιωματικούς από τον ΝΑΤΟ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της περίοδου αυτής συντοπίσαμε ότι δεν υπάρχει πλέον ένας συναγωνισμός ή ανταγωνισμός καλύτερα μεταξύ στρατιωτικών δομών Ευρωπαϊκής Ένωσης και στρατιωτικών δομών του ΝΑΤΟ. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ θετικό. Το ερώτημά μου όμως είναι το ακόλουθο. Εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η στρατιωτική συνεργασία με το ΝΑΤΟ και πώς επικοινωνείτε τελικά με τις δομές του ΝΑΤΟ. Έχετε ένα μόνιμο τακτικό διάβλο επικοινωνίας. Τι είδου σχέσεις αυτή τη στιγμή έχετε με τις δομές διοίκησης του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριος Γκάλερ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση που κάνατε για αυτόν τον γενικό απολογισμό του έργου του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας δίδεται κατά αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να κάνουμε κι εμείς κάποιες ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στο ρόλο εφαρμογή της παγκόσμια, στο ρόλο το δικό σα στην εφαρμογή τη παγκόσμια στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρχή τη εβδομάδα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ήρθε η ύπατη εκπρόσωπο Φεντερίκα Μογκερίνη και τη είπαμε θα μα παρουσιάσετε και στο μέλλον και άλλα σχέδια εφαρμογή τη παγκόσμια στρατηγική. Και θυμάμαι ότι μετά την Σύνοδο του 2013 είχε υποβάλει ένα κοινό έγγραφο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα και μα είχαν πει τότε αυτό το έγγραφο πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί. Εγώ τη ρώτησα τι γίνεται με, με το αρχικό αυτό έγγραφο αλλά δεν μου έχει δώσει ακόμα κάποια απάντηση. Επομένως το ερώτημά μου, η παράτησή μου είναι η ακόλουθη. Για άλλη μια φορά μιλάμε για ένα σχέδιο εφαρμογής, για ένα ακόμα σχέδιο εφαρμογής, ενώ δεν ξέρουμε καν τι γίνεται με τα προηγούμενα σχέδια τα οποία μας παρουσιάσατε στις αρχές του 2014. Εγώ ανέκαθεν έλεγα ότι όταν από τη μία πλευρά έχουμε το στρατηγικό προσανατολισμό της παγκόσμιας στρατηγικής θα πρέπει να το συνδυάζουμε με τις εξελίξεις των στρατιωτικών δυνατοτήτων μας. Θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη λευκή βίβλο για το ζήτημα αυτό. Και μόνο τότε θα καταφέρναμε να έχουμε και μια πραγματική έκθεση, αναθεώρηση αν θέλετε των αμυντικών μας ζητημάτων. Τότε μόνο θα γνωρίζαμε πραγματικά πού βρισκόμαστε και ποιες είναι δεσμεύσεις μπορούμε να πετύσουμε από τα κράτη-μέλη. Κάτι τέτοιο θα ήθελα εγώ να δω στο μέλλον. Επομένω, το ερώτημά μου είναι το ακόλουθο. Αν τυχόν κάποια στιγμή εγκρίνει μια τέτοια ιδέα η κυρία Μογκερίνη, είμαστε εμείς σε θέση να αρχίσουμε να συλλέγουμε πληροφορίες, στοιχεία, σχέδια από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερον, Προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και προσεκτικά για την ημέρα εκείνη που επιτέλους αποφασίσουν τα κράτη-μέλη να ενεργοποιήσουν το σύστημα ΠΕΣΚΟ, έχουμε αυτή τη στιγμή μία δυνατότητα μη στρατιωτικού σχεδιασμού και ικανοτήτων. Έχουμε το σχεδιασμό, τον έχουμε ενεργοποιήσει, αλλά δεν ασχολούμαστε καθόλου αυτή τη στιγμή με την ανάπτυξη των δυνάμεων. Αν λοιπόν δημιουργηθεί ένα μόνιμο στρατηγείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μόνιμο στρατιωτικό αρχηγείο, τότε θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποια στοιχεία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και ποιε δυνατότητε θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το στρατηγείο. Όταν ρώτησα την κυρία Φογκερίνη, μου είπε, Μογκερίνη μου πότε ότι αυτό εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Και εγώ τη είπα, μα εξαρτάται πραγματικά από εσά αυτό. Εσεί τουλάχιστον τροφοδοτείτε την κυρία Μογκερίνη με τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου τα κράτη-μέλη να ενθαρρυνθούν τελικά για να δημιουργήσουν το αρχηγείο αυτό. Και α μην ξεχνάμε ότι έχουμε και έναν νέο πρόεδρο πλέον στις ΗΠΑ, ο οποίο ε, για τον τομέα της ασφάλειας και της ε, άμυνας έχει μία πολιτική η οποία δεν είναι ακόμα απόλυτα προκαθορισμένη. Πήγε λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανασυνταχθούμε, να είμαστε προετοιμασμένοι και βασίζομαι σε εσά προκειμένου να καταφέρετε να δώσετε τα απαραίτητα στοιχεία στην κυρία Μογκερίνη για να ενθαρρυνθούν και τα κράτη-μέλη για να δημιουργήσουν αυτό το μόνιμο στρατιωτικό αρχηγείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενο ομιλητή. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Στρατηγέ. Στην αρχή της παρέμβασής σας είπατε ότι η διεθνής κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη σίγουρα αλλάζει συνεχώς και αλλάζει βέβαια και σήμερα. Από σήμερα αλλάζουν δραματικά και ολοκληρωτικά θα έλεγα οι προοπτικές που έχουμε. Ακριβώς όμως επειδή ε, μεταβάλλεται συνεχώς η κατάσταση, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες. Ενδεχομένως ε, να μην ε, αρέσκονται οι στρατιώτες του να απαντούν πολιτικά ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε κάπως για τις προτεραιότητες αυτές που θα πρέπει να έχουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρουσία μας στην Σομαλία, η παρουσία μας στο Μαλί, η παρουσία μας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι πάρα πολύ σημαντική από ανθρωπιστικής πλευράς. Οι επιχειρήσεις όμως αυτές απλώς επιβεβαιώνουν, θεωρώ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και είναι σε θέση να συμμετέχει σε μεγαλεπίβολες τέτοιες επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να καταφέρνουμε να καλύπτουμε και τις δεσμεύσεις μας απέντη στα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες και αναφέρομαι εδώ πέρα στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Πριν από 4-5 χρόνια, George Frisbane έγραψε ένα δοκίμιο για την ε, σχετικότητα της, ε, του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά διερωτήθηκε αν πρόκειται για μια στρατιωτική συμμαχία, για μια πολιτική συμμαχία. Νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει εμείς μέσω συγκεκριμένων δράσεων να δείξουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν ισχύει μια τέτοια αμφισημία. Να σας δώσω ένα ακόμα παράδειγμα. Αναφέρομαι στην περιοχή της Μεσογείου. Εδώ και δέκα ολόκληρους μήνες βλέπουμε ότι έχουν αναλυφθεί δεσμεύσεις οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί όσον αφορά την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών. Υποτίθεται ότι έχουμε εκεί πέρα μια εκτοφυλακή, υποτίθεται ότι έχουμε επιτόπου στρατιώτες για να πατάξουν αυτό το φαινόμενο. Αν δεν ήταν εκεί πέρα, το φαινόμενο αυτό θα γνώριζε όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Πριν από 1,5 χρόνο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσημα αποφάσισε να καταπολεμήσει τα δίκτυα διακινητών προσφύγων και μεταναστών στις ακτές των χωρών προέλευσης. Λίγο αργότερα μας είπαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει, μάλλον θα έπρεπε να γίνει βάσει διπλωματικής εντολής. Δόθηκε η διπλωματική αυτή εντολή με περιορισμένο βέβαια πεδίο εφαρμογή. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε συμβάλει τότε πάρα πολύ στο να εγκριθεί η συμφωνία αυτή. Πώς θα μπορούσε όμως να ευοδοθεί μια τέτοια επιχείρηση και στο μέλλον. Η επιχείρηση Σοφία είναι πολύ σημαντική, η ανθρωπιστική, ανθρωπιστική της διάσταση είναι πολύ σημαντική, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί, να είναι αποτελεσματική τελικά επιχείρηση αυτή και όντω να συμβάλλει στην πάταξη των δικτύων αυτών. Τέλος, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, ποιες έχετε εντοπίσει εσείς ως σημαντικότερες προκλήσεις, σε ποιες θα πρέπει να εστιαστούμε, ποιες απειλές μπορούμε τελικά να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε. Αν θα καταφέρουμε να εντοπίσουμε λοιπόν τις προτεραιότητές μας, θα βρεθούμε σε πολύ δεινή κατάσταση. Ξέρετε, τον Ντεγκόλ μιλούσε για μια πραγματική παρουσία, να έχει κανείς μια πραγματική, να είναι πραγματικά προβεβλημένος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ως Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε προβεβλημένοι μέσω της δράσης μας στο παγκόσμιο προσκήνιο. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να εντοπίσουμε συγκεκριμένα καθήκοντα και συγκεκριμένες προτεραιότητες. Ποιες λοιπόν είναι κατ' εσάς οι σημαντικότερες προκλήσεις, πού πρέπει να εστιαστούμε. πού θα πρέπει να συμπληρώνουμε τη δράση του ΝΑΤΟ, πού θα πρέπει να αναλάβουμε εμεί τη δική μας πρωτοβουλία. Και προφανώς δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέλη του ΝΑΤΟ, ορισμένα διατηρούν ουδέτερη στάση, αλλά συνεργαζόμαστε όλοι μας. Η κυρία Λέζινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ορισμένες ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις η, σφαιρική, η παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, περιλαμβάνει μια προσαρμογή του μεγέθους των στρατευμάτων. Ε, μέχρι στιγμής ορίζονται στον αριθμό 60.000. Ε, είναι αναγκαία λοιπόν μια προσαρμογή του headline goal εδώ, τους, και αν ναι, μέχρι σε ποιο αριθμό. Ε, τα στρατικοί προπολογισμοί των χωρών είναι 200 δις ευρώ ανά έτος. Πώς αξιολογείται το επιπλέον ανάγκη επένδυσης προκειμένου να εφαρμοστεί η παγκόσμια στρατηγική, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική υπηρεσία του γερμανικού Bundestag πριν από λίγο καιρό δημοσίευσε μία γνωμάτευση στην οποία αναφέρεται το εξή. Η Γερμανία ε, ενδεχομένως ε, θα μπορούσε ε, να καλύψει την θέση του Γενικού Διευθυντή του Στρατιωτικού Προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά, μετά το Brexit. Ευχαριστώ για την τελευταία παρέμβαση για αυτή τη συζήτηση. Οπότε, στρατηγία, αν μπορείτε, απαντήστε στις ε, ερωτήσεις και τις ε, παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. κάπως με καθησυχάζουν. Οι ερωτήσεις σας που ήταν τόσο εύστοχες γιατί σημαίνει ότι παίρνετε την υπόθεση αυτή στα σοβαρά. Μπράβο σας. Τώρα, όσον αφορά τον ΝΑΤΟ, έχουμε τις σχετικές δυνάμεις και 90% αποτελούν δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Οπότε υπάρχει διαλειτουργικότητα πλήρω με το ΝΑΤΟ όσον αφορά το προσωπικό της Ένωσης. Και στο καθημερινό έργο μας, σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, αυτή η διαλειτουργικότητα αυξάνεται, βελτιώνεται. Εδώ και χρόνια επιχειρούμε και σε λειτουργικό επίπεδο και κατά θάλασσα έχουμε κοινή δράση. Γιατί και εκεί συνεργαζόμαστε με τον ΝΑΤΟ και στην Μεσόγειο. Τώρα αυτό το δικό μου επιτελείο και το δικό μου ρόλο. Έχω τακτές επαφές με το στατικό προσωπικό του ΝΑΤΟ και τουλάχιστον μία φορά το μήνα συναντιόμεθα με τον Γενικό Διευθυντή και έχουμε επομένω ε, επαφέ με του ομολόγου μα, το προσωπικό του ΝΑΤΟ, ανταλλαγή πληροφοριών. Συστάμε ό,τι πρόβλημα προκύπτει. Έχουμε ένα πολιτικό πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα και μας περιορίζει, οπότε δεν μπορούμε από στρατηγική πλευρά να ε, δράσουμε όσο θα θέλαμε σε βάθο. Αλλά αυτή είναι η πολιτική συγκυρία και από πλευρά τη ΝΑΤΟ και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι τόσο ευχάριστο από τη μα πλευρά. Αλλά τι να κάνουμε. Τόσο αφορά την πρακτική συνεργασία, μπορούμε να ασχοληθούμε εις βάθος με τα θέματα, αλλά πάντοτε υπάρχει ένα όριο Οπότε και θα πρέπει να αναφερθούμε ε, στους ε, πολιτικούς ε, και έτσι να εξασφαλιστεί κάποια συνέχεια στην πολιτική συνεργασία. Επομένω, υπάρχει κατανόηση πλήρη σε στρατηγικό επίπεδο, υπάρχει αγαστή συνεργασία. Και όσο είναι δυνατόν, συνεργαζόμαστε με τον ΝΑΤΟ. Είναι ενιαίες οι δυνάμεις του κάθε κράτους μέλους. Υπάρχει αντιστοιχεία κράτων, κράτων μελών της Ένωσης και του, και του, των μελών του ΝΑΤΟ. Όπως είπαμε, επομένω, είναι ψηλά πήγε στη πλευρά και τα όρια είναι δεδομένα όσον αφορά την πολιτική πτυχή της εργασίας. Τώρα για την γενικότερη σφαιρική στρατηγική. Υπολήθηκε κάποια ερώτηση για την απόφαση του Συμβουλίου του 2013 και τόσο αφορούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Μήνας. Από πλευρά ε, δυνατοτήτων και δυναμικού η δυσκολία είναι στο ότι αφενός τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν τη θέληση να προβούν σε προμήθειες, σε διαγωνισμούς κοινούς και πολλά χρόνια αυτό ήταν ένα θέμα. Το πώς θα πείσουμε τα κατημέλια να ασχοληθούν και να συμμορφωθούν με το θέμα αυτό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα που είναι ένα φορέας, ένα όργανο το οποίο βοηθά τα κράτη-μέλη. Το θέμα μόνο λοιπόν, είναι όμω να υπάρχει βούληση των κρατών μελών που δεν είναι δεδομένη, ούτε τόσο έντονη. Τα πράγματα είναι πιο ρόδινα τώρα σχετικά με αυτό. Γιατί έχουμε τι στρατηγικέ κατευθυντήρε γραμμέ. υπάρχει περισσότερη κατανόηση ο πλευρά Ότι κανεί δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο του και ότι εν οι ενώση δύναμη. Όμω γίνονται πολλά σε περιφερειακό επίπεδο. Δημερό, τριμερό. Ακόμα και πολυμερός. Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ ή στα πλαίσια άλλων δομών και ρυθμίσεων περιφερειακών. Ας πούμε σε σχέση με τη Σκανδιναβική Συμφωνία μήνες. Βεβαίως είναι και θέμα αμυντικής βιομηχανίας. και το τι όρθιση δίνεται από την αγορά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από αυτές τις μεταβλές εξαρτάται το πόσο εις βάθος μπορούμε να δράσουμε τώρα όσον αφορά το δυναμικό, τις δυνατότητες, πώς βλέπουμε τα πράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε από στρατιωτικής πλευράς. Έχουμε τον κατάλογο απαιτουμένων ή προαπαιτουμένων 05. Θα πρέπει πρώτα απ' να γίνει μια αξιολόγηση επί τη βάση κατευθυντηρίων πολιτικών των κρατών μελών. Να εγκρίνουν το πλάνο υλοποίηση. Να δούμε τι προτεραιότητε, τι φιλοδοξίε έχουμε, τι γίνεται με τι επιχειρήσει, τι στρατιωτικέ, τι γίνεται με τι πολιτικέ ε, αποστολέ. Οπότε ρωτούμε και νέα σενάρια για να δούμε κατά πόσον αυτά τα προπετούμενα προϋποθέσεις έχουν αλλάξει ή όχι. για να πώς αυτά συμβαδίζουν με τα όσα ζητεί ως προποθέσεις έχει η τάξη η υπηρεσία άμυνας. Ακόμα δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο κατά πόσο θα πρέπει να θεωρήσουμε κάποιο τίτλο, κάποιο κεφάλαιο προς το παρόν και να κάνουμε ένα άλλο προγραμματισμό. Τώρα, όσο αφορά τη συνεργασία των διαφορετικών δομών μας, το τι είναι, αιτία ή μέσον για να καταφέρουμε κάτι. Αλλά πάντως έτσι μπορούσαμε να επιταχύνουμε την εξέλιξη όσο αφορά συνεργασία για τα θέματα της άμυνας. Πάντως και από αυτού τα κρατημέλη έχουν το πάνω χέρι πρέπει να αποφασίσουν τώρα. Τώρα όσον αφορά το CPCC το Civilian Planning και Conduct Capability. Να δούμε τι γίνεται από πλευράς πολιτικών αποστολών και επιχειρήσεων. Χρειάζεται πάντοτε να συνοδεύονται αυτή η προσπάθεια και με στρατιωτική υποστήριξη. Χρειάζεται κάποια συνέργεια Υπάρχουν επίσης και οι αποστολές ε, εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Πάντως, είμαι βόρειος και εμείς οι βόρειοι είμαστε ρεαλιστές. Και θεωρώ ότι θα πρέπει ο προσύγγι να γίνεται βήμα-βήμα. Να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε σήμερα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα με τους σημερινούς πόρους. να γίνει το αυτοκίνητο τουρμποκίνητο. Και σύμφωνα το Συμβουλίου μετά να δούμε τι μπορούμε να θεωρήσουμε το πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα και να δούμε μετά τα νομικά θέματα τα οποία παίρνουν χρόνο για να επιληθούν. Άρα θα πρέπει έτσι να κινηθούμε, όπως είπαμε, βήμα-βήμα. και σε επίπεδο υπάτης εκπροσώπου να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν και τι ευκαιρίες υπάρχουν τώρα για τις προτεραιότητες. Η κυρία Μογκερίνη έχει χαράξει κάποιο, κάποιο προτεραιότητες, έχει βάλει τον πύχη των φιλοδοξιών μας και για στρατιωτικές επιχειρήσεις και για πολιτικές αποστολές και εκτός συνόρων διάφορα είδη αποστολών για συνεργασίες, εταιρικέ σχέσεις τη συνεργασία με διάφορους μια που μόνοι μας δεν μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα το ΝΑΤΟ, Αφρικανική Ένωση αυτούς τους εταίρους και άλλους αλλά επίσης και την οικοδόμηση δυνατοτήτων. Για τις τρίτες χώρες. Άρα θα δώσουμε επιπληκτική βοήθεια στις χώρες εκείνες. Όμως χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ανάπτυξη. Άρα, αυτή είναι η αφιτερία, το θεμέλιο του έργου μας. την ίδια ότι κάνουμε εκτός συνόρων βοηθά και στην ασφάλεια της Ευρώπης. Άλλη βέβαια είναι η προστασία της Ευρώπης. Υπήρξαν παρεξηγήσεις στο πρόσφατο παρελθόν σε σχέση με αυτό. Να δούμε τώρα τα θέματα των οργανισμών το ΝΑΤΟ κατά κάποιο τρόπο έχει γυρίσει στις απαρχές σύμφωνα με το άρθρο 5 δηλαδή το πώ θα γίνει η συλλογική άμυνα και αυτό το βλέπετε και από την ευξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ τώρα προς Ανατολάς και Βορειοανατολικά σε εκείνα τα κράτη-μέλη. Επίσης, το ΝΑΤΟ συμβάλλει σε επιχειρήσεις και αποστολές στο εξωτερικό. αλλά δεν καλύπτει να δυνατότητες του ΝΑΤΟ δηλαδή το άρθρο 5 και όσον αφορά την προστασία της ε, Ευρώπης εκεί υπάρχουν πολλά περιθώρια γιατί έχουμε ε, την παράνομη δρανάστευση, έχουμε την τρομοκρατία, έχουμε το εμπόριο ανθρώπων, το, την εμπορία. έχουμε το κυβέρνο έγκλημα. Πολλά θέματα τα οποία δημιουργούν πάρα πολύ υλικό είναι καλύτερα και μικρότερα προβλήματα και από θεσμική πλευρά, όλα αυτά έχουν σχέση και καλύπτονται από τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόκειται μα για προστασία Ευρωπαίων και Ευρωπαϊκού Εδάφου, ευρωπαϊκή Επικράτηση. Αυτό θα πρέπει με προσοχή να μα απασχολήσει για την προστασία των συνόρων μας σημαίνει ότι θέλουμε να αποτρέψουμε τους τρομοκράτες να έρχονται στην Ευρώπη και έτσι θα βοηθήσουμε στην ασφάλεια και προστασία των πολιτών. Οπότε βέβαια εκεί έχουμε κάποια όρια. Τα όρια της ε, κοινή πολιτικής, ε, άμυνας και ασφάλειας. Έχουμε επίσης και τη ρήτρα ελληνικής, σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε εντός και τι εκτός συνόρων. Οπότε και εδώ το μπαλάκι είναι στο γήπεδο των κρατών μελών για το ποιες αρχές θα δράσουν από αυτού. Χωροφυλακή, αστυνομία, τέτοιου είδους διοκτικές αρχές. Στη Μεσόγειο έχουμε την επιχείρηση Σοφία. Έχει όρια και περιορισμού αυτή η επιχείρηση. Πολύ σωστά τα είπατε. Έχουμε όλες αυτές τις διασώσεις, μιλάμε για πάνω από 32.000 ε, ε, πολιτών από τις ε, τρίτες χώρες. Πρόκειται για μια προσπάθεια ανθρωπιστική. βοηθάει βέβαια και εκτός από τη διάσωση και το να διαλύσουμε τα δίκτυα των ε, διακινητών, με κάθε μέσο να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τα σύνορα στη Μεσόγειο. Μόνο εμείς μπορούμε να το δούμε, μόνο εμείς έχουμε τα μέσα προς τούτο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αόρια σε αυτή την εντολή που έχουμε. Και αυτό είναι και δυσκολία. Θα πρέπει να δράσουμε εκτός της ε, λιβικής υφαλοκρηπίδας και εναερίου χώρου. Στην αρχή θεωρούσαμε ότι θα πάμε να δράσουμε εκεί όταν υπήρχε η εντολή, αλλά έτσι όπω έγιναν τα πράγματα, το τώρα που κατέληξε η Λιβύη να είναι ένα χρεοκοπημένο κράτο και οπότε μα ζήτησε η διακυβέρνηση να πάει εκεί μια που βρίσκεται είναι εμφυλίο. Άρα τα πράγματα δυσκολεύουν όλο και περισσότερο. Και για να προσπαθήσουμε κάτι να κάνουμε, πήρε την εντολή η επιχείρηση Σοφία, ούτω ώστε να αρχίσουν να βοηθούν την ακτοφυλακή της χώρας εκείνης, της Λιβύης, εκπαιδευτικές δράσεις τελείο Οκτωβρίου και έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις ελληνικές αρχές για τους ανθρώπινους πόρους να τους δώσουμε κάποιες δυνατότητες ε, κατά θάλασσα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σύνορά τους. Έτσι μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, έτσι ίσως ε, δυσκολέψουμε τους ε, διακινητές. Γιατί ε, τη σήμερα ημέρα τα πάνε μια χαρά έχουν εύκολο έργο. Βέβαια εξαρτάται και οι πολιτικοί τι αποφασίζουν για κάθε φάση των στρατηγικών επιχειρήσεων. Αλλά φροντίζοντας την υπόθεση της ασφάλειας σε Μεσόγειο και Λιβικές ακτές αυτό δεν είναι το γενικότερο πρόβλημα γιατί υπάρχουν πολλές αιτίε των προβλημάτων και αυτές οι αιτίε βρίσκονται και στην Αφρική οπότε έχουμε και εκεί πέρα κάποιο είδους ε, επιχειρήσεις και αποστολές που πολλοί λένε ότι είναι σταγόνο το ωκεανό εγώ διαφωνώ θα πρέπει να δούμε πώς θα αναβαθμίσουν την ασφάλεια στις χώρες που πρέπει. Και πρέπει να βοηθήσουμε και να λάβουν και το ρόλο που πρέπει αυτές οι χώρες για τον εαυτό τους. Και αυτό θα τα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της, αλλά θα τα κάνει σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και την Αφρικανική Ένωση. Δεν είναι θέμα θεσμικό, δεν είναι θέμα φθόνου προς τον ΝΑΤΟ. Είναι θέμα κοινού σκοπού, κοινών απειλών. Αλλά δεν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού με τον ΝΑΤΟ. Όχι, δεν είμαστε ανταγωνιστές του ΝΑΤΟ. Είμαστε ε, συνεργάτες, εταίροι. Όσον αφορά τώρα το θέμα των χρημάτων που χρειαζόμαστε, είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Αλλά θα έλεγα ότι θεωρητικά η κατανομή των κονδυλίων στις χώρες μέλη, έχοντας κατά νου ότι ο προϋπολογισμός αυξάνεται ελαφρά. Εάν οι χώρες μέλη χρησιμοποιήσουν έξυπνο τρόπο τον προπολογισμό τους, θα μπορούμε να έχουμε αρκετά κονδύλια, καρδιά χρήματα για τις επενδύσεις. Αλλά το να γίνει έξυπνα η επένδυση σημαίνει να, γίνει από ε, να γίνουν από κοινού οι επενδύσεις. Ε, ε, θα πρέπει οι χώρες μέλη να συνεργαστούν γιατί δεν υπάρχουν πολλά θέματα ε, τα οποία είναι κυρίως ε, εθνικά. Συνήθως είναι, αφορούν όλες τις χώρες. Ε, θυμηθείτε ότι και 28 χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Ε, και είναι καλό να χρησιμοποιηθεί ο, το, να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των χωρών ε, μελών. Είναι κρίσιμες αυτές οι επενδύσεις όσον αφορά την αύξηση του δυναμικού μας. Δεν υπάρχουν αριθμοί ακριβώς. Και αν η επένδυση των χρημάτων γίνει περισσότερο για τα πολυεθνικά ε, προγράμματα, αυτό θα είναι ε, χρήσιμο, θα είναι πιο έξυπνο. Γιατί υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία αφορούν πολλές χώρες. Όσον αφορά το Brexit, το άρθρο 50 δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί ε, και αυτό θα περιοδοτούσε τις εξελίξεις. Εγώ θα έπαιρνα μια αμυντική ε, θέση γιατί ε, έχω στο προσωπικό μου 15 Βρετανούς όλοι αυτοί είναι 100% υπέρ της Ευρώπης είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι και θέλουν να, εισβάλ, να συνεισφέρουν όσο περισσότερο μπορούν ε, στην Ευρώπη. Δεν ξέρουμε ποιες ακριβώς θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι έχουμε ακόμα ανάμεσά μας αυτούς τους ανθρώπους, τους Βρετανούς, οι οποίοι ε, συνεισφέρουν ε, Δεν είναι πολλά τα 15 αυτά πρόσωπα, αλλά εάν ε, θέλαμε να τα αντικαταστήσουμε με ανθρώπους από άλλες χώρες, νομίζω ότι θα υπήρχαν δυσκολίες. Στην περίπτωση του Ενωμένου Βασιλείου, θα έλεγα ότι είναι μια ισχυρή, αν όχι ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη και αν όντως συμβεί το Brexit, αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο δυναμικό μας. Αν το δούμε καθαρά στρατιωτικά, θα ήταν πολύ ωφέλιμο να συνεχίσουμε να έχουμε τη Μεγάλη Βρετανία ε, έστω και αν γίνει το Brexit. Η Μεγάλη Βρετανία θα παραμείνει μια ευρωπαϊκή δύναμη, γιατί οι κίνδυνοι ε, παραμένουν οι ίδιοι, είτε με Brexit είτε χωρίς. Κύριε Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την ιδιαίτερα αυτή ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Ελπίζουμε να έρθετε πάλι σύντομα στην Επιτροπή μας ε, για να μας για τις ε, περαιτέρω εξελίξεις που θα έχουμε. Διανύουμε ενδιαφέροντες καιρούς. Σας ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά πολύ και προσβλέπουμε στην επόμενη παρέμβασή σας εδώ στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μείνετε όμως σας παρακαλώ πολύ γιατί έχουμε ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον σημείο στη μερίσια διάταξη. Uh, well, Κυρίες και κύριοι, ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο πρέσβης του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το υποεξέταση ζήτημα έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Διατλαντική συνεργασία για την ασφάλεια. Θα θέλαμε λοιπόν μαζί σας, κύριε πρέσβη, να συζητήσουμε την καναδική προοπτική όσον αφορά τη διατλαντική συνεργασία για την ασφάλεια. Ήθιστε κάθε φορά που μιλάμε για διατλαντική συνεργασία για την ασφάλεια να αναφερόμαστε κυρίως στη σχέση που έχουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Είτε σε διμερές, είτε σε πολυμερές επίπεδο, είτε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. και συχνά ξεχνάμε την της συμβολή του άλλου σημαντικού μας εταίρου της Βορείου Αμερικής, δηλαδή τη συμβολή του Καναδά. Η σχέση λοιπόν αυτή είναι μακροχρόνια. Βλέπω ότι φοράτε και την παπαρούνα. Πράγμα που μου θυμίζει την τεράστια συμβολή των Καναδών τον προηγούμενο αιώνα, κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για την ε, διασφάλιση της ε, ειρήνης στην Ευρώπη και όλες αυτές τις θυσίες που έκαναν οι πολίτες του Καναδά. Εξοχότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, έστω και μια προχωρημένη ώρα στην Επιτροπή μας. Έχετε ευθύ αμέσω το λόγο. Πρόκειται προφανώ για τον κύριο Ντάνιελ Κοστέλο, πρέσβη του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ που παραμείνατε εδώ στην αίθουσα αυτή μετά από μια πολύ μεγάλη ημέρα. Σας ευχαριστώ επίσης επειδή αναγνωρίζετε το ρόλο του Καναδά στη Διατλαντική Συνεργασία για την Ασφάλεια. Μα ξεχνάτε πολύ συχνά, θα συνεχίσουμε να λέμε εμεί ότι δεν θέλουμε όμω να μα ξεχνάτε, επιθυμούμε να μα αναγνωρίζετε ω σημαντικό εταίρο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που αναγνωρίζετε επίση το ρόλο του Καναδά στην διασφάλιση τη ειρήνη στην Ευρώπη κατά τον προηγούμενο αιώνα. Είναι μια εβδομάδα που ξέρω τη φορά με το λουλούδι αυτό, την Παπαρούνα, προ υπενθύμηση τη συμβολή του Καναδά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα μιλήσω καταρχά στα γαλλικά. Θα κάνω μια παρουσίαση στα αγγλικά σύντομη παρουσίαση, σας το υπόσχομαι. Αλλά ξέρετε ότι στον Καναδά χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε και τη γλώσσα του Μολιέρου. Θα μιλήσω όμως τώρα αγγλικά. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί ήταν πολύ μεγάλη μέρα για σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μιλήσω για τη διατλαντική συνεργασία για την ασφάλεια και για τη συμβολή του Καναδά. Θα έλεγα πολύ σύντομα ότι ε, έχουμε κοινέ διεθνείς προτεραιότητες και αυτό δεν είναι τυχαίο. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα για κάποιους βασικούς τομείς τους οποίους εμπλεκόμαστε δυναμικά από κοινού. Και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και την διμερή σχέση και συνεργασία μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε και ποιες είναι οι μελλοντικές μας προοπτικές. Νομίζω ότι θα είμαι πολύ σύντομος γιατί προτιμώ να ακούσω τις δικές σας παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας εταίρος εκ των ουκάνευ. Μια δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί στην δυνατό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμεριζόμαστε κοινέ θεμελιώδεις αξίες. Γιορτάζουμε την 40η επέτειο των επίσημων διμερών μας σχέσεων, αλλά όπως είπε και η πρόοδος, έχουμε μια πολύ μακροχρόνια ιστορία. Ήμασταν πάντα στο πλευρό της Ευρώπης και αυτό αποδεικνύεται και από την ιστορία την Όσον αφορά τώρα τις διεθνείς μας προτεραιότητες, βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόλυτη ευθυγράμμιση μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε και εμείς διεθνή σταθερότητα και ειρήνη, ιδίως στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θερώ, αναφέρομαι εδώ πέρα στην ε, ανατολική πλευρά, στην νότια πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρομαι στη Μέση Ανατολή, στην καταπολέμηση τρομοκρατίας, στην καταπολέμηση της ρίζος παστικοποίησης. Θέλουμε να προωθήσουμε την ειρήνη για τον πλουραλισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού στον κόσμο. Δεσμευόμαστε επίσης για τα πολυμερή πλαίσια, την ενίσχυση των πολυμερών σχέσεων, την ενίσχυση του πολυμερισμού, τη χρηστή παγκόσμια κυβέρνηση και Δεσμευόμαστε πάρα πολύ για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, ιδίως την αυτή προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε του νέου στόχου βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων εθνών και θέλουμε να αναλάβουμε δράση τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά για την αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή και για τη μετάβαση προ πιο καθαρέ πηγέ ενέργεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επενδύουμε επίση σε ανοιχτέ κοινωνίε, σε μια οικονομική ανάπτυξη χωρί αποκλεισμού και στο εσωτερικό του Καναδά και με όλου του εμπορικού μα και οικονομικού εταίρου. Πριν από μία μισή εβδομάδα ο Πρωθυπουργό τη χώρα μου ήταν στι Βρυξέλλε και υπέγραψε καταρχά συμφωνία ΣΕΤΑ που θα τεθεί πολύ σύντομα σε ισχύ, καθώ επίση και την συμφωνία στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά. Και οι δύο αυτέ συμφωνίε τονίζουν τι κοινέ μα θεμελιώδει αξίε και νομίζω ότι θα μα επιτρέψουν τελικά να φέρουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο εγκύτητα και συνεργασία τη μακροχρόνια σχέση που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίω αν δούμε τη νέα παγκόσμια στρατηγική που ανακοίνωσε πριν από μερικέ μέρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίση να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι οι διεθνεί αυτές προτεραιότητες είναι προτεραιότητες τόσο του Καναδά όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι τυχαίο αυτό ακριβώς επειδή έχουμε κοινέ αξίε, όπως σα είπα, δεσμευόμαστε για τις αξίες αυτές, θεωρούμε ότι είναι προ το κοινό μα συμφέρον να τις προασπίσουμε και προφανώς η δική μα ασφάλεια συνδέεται με τη δική σα την ασφάλεια, η δική μα ευημερία συνδέεται με μια ευημερούσα Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορά λοιπόν που κοιτάμε τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνειδητοποιούμε ότι οι προκλήσεις αυτέ είναι και δικέ μα προκλήσει και καλούμεθα και εμεί να τι αντιμετωπίσουμε. Να σα δώσω κάποια παραδείγματα. Πρώτον, συνασπισμό κατά του Ισλαμικού κράτου. Ήδη από την αρχή είχαμε δεσμευτεί ω χώρα στι προσπάθειε τη συμμαχία που ξεκίνησαν το 2014. Συμμετέχουμε και στι πέντε γραμμέ τι επιχειρησιακέ έχουμε μια σημαντική στρατιωτική παρουσία επιτόπου. Συμμετείχαμε επίσης στις αεροπορικές, ε, ε, αεροπορικούς βανδρισμούς που γίνανε τόσο στο Ιράκ και στη Συρία. Έχουμε τριπλασιάσει την ενίσχυσή μας όσον αφορά τη δημιουργία επιτόπιων στρατιωτικών δυνάμεων. 300 Καναδοί είναι παρόντες επιτόπου και συμβάλλουν πάρα πολύ στην υποστήριξη των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράκ. ...1,6 δισεκατομμύριο δολάρια πρόκειται να δώσουμε τα επόμενα τρία χρόνια... ...στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης περιφερειακής ανταπόκρισης για τη Συρία και το Ιράκ... ...για ζητήματα ασφάλειας και ζητήματα σταθεροποίησης, ανάπτυξης και σχεδιασμό ανθρωπιστικής βοήθειας και επίσης είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι διπλωματικά στην Ηνωμένα Έθνη και στο διεθνές, στη Διεθνή Ομάδα υποστήριξη για τη Συρία, καθώς επίσης και σε άλλα διεθνή φόρουμ, με απότερο στόχο να καταφέρουμε να επιφέρουμε μια ειρηνική λύση στην απέσει αυτή η ανθρωπιστική καταστροφή την οποία βλέπουμε στην Συρία. Εδώ και πάρα πολύ καιρό θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθεί δράση από την ΟΕΕ προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στο Χαλέπι, ιδίως όσον αφορά την ανθρωπιστική πλευρά της ε, καταστροφής. Αν δούμε τώρα πέρα από το μεσανατολικό και τα ιδιαίτερα πιεστικά προβλήματα που έχουμε εκεί, θα μπορούσα να αφαιρθώ στην ανατολική εταιρική σχέση. Σας είπα ότι ανέκαθεν υποστηρίζαμε την Ουκρανία. 1,3 Καναδοί είναι ουκρανικής καταγωγής και έχουμε και πάρα πολλούς άλλους Καναδούς πολίτες που κατάγονται από την Ανατολική Ευρώπη έχουμε διατηρήσει αμετάκλητη την τοποθέτησή μας ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την τωρινή κατάσταση της Ουκρανίας και θα πρέπει προφανώς να ισχύουν οι κυρώσεις αυτές μέχρι να αρχίσουν να εφαρμόζονται πλήρως οι συμφωνίες του Μίνσκα. Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα έλεγα ότι από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις του Euromaidan και μετά και ιδίω με την προσάρτηση της Κρυμαίας αναλάβαμε δράση όχι μόνο στα πλαίσια των κυρώσεων αλλά δώσαμε και 700 εκατομμύρια δολάρια σε τεχνοοικονομική υποστήριξη Στέλναμε επίσης επιτηρητές ε, των τοπικών εκλογών και σε διμερές επίπεδο δεσμευτήκαμε, δεσμεύσαμε μισό εκατομμύρια δολάρια που θα πάρουν τη μορφή τεχνικής υποστήριξης προς την Ουκρανία και έχουμε 200 στρατιωτικούς ε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Ουκρανία προκειμένου να συμβάλλουν στην οικοδόμηση στρατιωτικών δυνατοτήτων στον Καναδά και να συμβάλλουν επίσης στην κατάρτιση του εκεί στρατιωτικού προσωπικού. Να ενταφερθώ επίσης και σε ένα άλλο τομέα, στο ΝΑΤΟ. Ξέρετε ότι ο Καναδάς είναι από τα μέλη του, του ΝΑΤΟ. Θεωρούμε ότι το ΝΑΤΟ είναι μια πολύ σημαντική πολιτική και στρατηγική σημασία, θεμελιώδους ιστορική σημασίας. Συμβάλαμε λοιπόν στην ίδρυση του ΝΑΤΟ πριν από 65 χρόνια και γι' αυτό ακριβώς το λόγο συμμετείχαμε ανέκαθεν ιδιαίτερα δραστήρια και συμμετέχουμε βέβαια σε αποστολές και επιχειρήσεις στο Αφγανιστά, στην Λιβύη, Ανήκουμε επίσης στην μονάδα εκείνη του ΝΑΤΟ που είχε να κάνει με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των δικτύων διακινητών στη Μεσόγειο και έχουμε παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη, κυρίως μέσα σε προγράμματα κατάρτισης. Ο Πρωθυπουργό Τρουντό ανέφερε στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Βαρσοβία ότι ο Καναδάς θα είναι μία από τις πιο δραστήριες χώρες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ προκειμένου να έχουμε μια πιο αποτελεσματική διεξαγωγή των ε, μονάδων μάχης, ενεργοποίηση μάλλον των μονάδων μάχης σε, διάφορα, ε, σε διάφορες ε, περιοχές του κόσμου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να στέλνουμε τόσο αεροσκάφη όσο και φρεγάτες στις περιοχές εκείνες όπου έχουμε αποστολές του ΝΑΤΟ. Είναι πάρα πολύ σημαντική θεωρώ συμμετοχή μας αυτή γιατί αυξάνει τόσο την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ όσο και τις προσπάθειες αποτροπής των συγκρούσεων. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συνεργασία μεταξύ πολύ για την κοινή δήλωση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την κοινή δήλωση μεταξύ ευρωπαικη ενωση και ΝΑΤΟ που είδαμε πέρυσι στην Βαρσοβία και θέλουμε το στομότερο δυνατό να υλοποιηθούν οι προτεραιοτητε που βρίσκουμε στη δήλωση αυτή, οπω για παράδειγμα η καταπολέμηση τη εγκληματικοτητα στο διαδίκτυο ή η ανάληψη κοινή δράση σε αλλου τομει μεταξύ ευρωπαικη ενωση και ΝΑΤΟ. Είμαστε υπέρ τη φιλοδοξια ευρωπαικη ενωση για την αύξηση της συνεργασίας για την πολιτική άμυνας και ασφάλειας και σε συνεργασία βέβαια με το ΝΑΤΟ. Τώρα σε διμερές επίπεδο να αναφέρω δύο πράγματα, δύο στοιχεία της διμερούς μας συνεργασίας που δεν τα γνωρίζετε οι περισσότεροι. Θεωρώ ότι είμαστε ο πιο σημαντικός μη ευρωπαϊκός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις αποστολές ΚΕΠΑ και όσον αφορά τις αποστολές επιτήρησης εκλογών σε 20 εκλογές ήμασταν παρόντες στην Αφρική, την Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές του κόσμου και είμαστε πάντα στο πλευρό των επιτηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς επειδή έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με εσά, μπορέσαμε να πάμε κι εμείς ως Καναδάς, ως Επιτροπή Επιτήρηση των Εκλογών από τον Καναδά, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Θα θέλαμε να συνεχιστεί αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τις αποστολές ΚΕΠΑ. Συμμετείχαμε, νομίζω, περισσότερο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 10 από τις 34 αποστολές και έπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αρχίσει να ισχύουν από το 2003. Η δική μας συμβολή ήταν κυρίως κατάρτιση αστυνομικών δυνάμεων και στρατιωτικών δυνάμεων και έχουμε καταφέρει να συμβάλλουμε όχι μόνο με εξοπλισμό αλλά και χρηματοδοτικά στο Μαλί, στο Κονγκό, στην πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, στη Βοσνία, στο Αφγανιστάν, στο Κωσυφοπαίδιο και έχουμε δύο αποστολέ αυτή τη στιγμή, υποστήριξη τη Ουκρανία και υποστήριξη τη δυτική όχθη με τη συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε να επεκταθεί η συνεργασία μα αυτή, αλλά αυτή τη στιγμή στον Καναδά προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά σε αποστολές ειρήνευσης και σταθεροποίηση. Ακόμα και αν μερικές φορές δίδεται η εντύπωση ότι έχουμε κυρίως συγκρούσεις και αστάθεια σε διάφορες περιοχές του κόσμου, θεωρώ ότι η κατάσταση τελικά ε, διαφοροποιείται. Δεν νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε τόσο πολύ με αντιπαραθέσεις και πολέμους μεταξύ κρατών, αλλά περισσότερο με εξεγέρσεις ή τρομοκρατικές δραστηριότητες. Πρέπει λοιπόν να αναπροσαρμόσουμε κι εμείς τη δική μας τη δράση, προκειμένου να προασπίσουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε αλυσίδα αξιών, να καταφέρουμε δηλαδή να ενισχύσουμε την ειρήνη, να μετριάσουμε τις συγκρούσεις και να επανοικοδομήσουμε τις κοινωνίες οι οποίες βγαίνουν από συγκρούσεις. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνησή μου ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα 450 εκατομμυρίων ευρώ επιχειρήσεις ε, οικοδόμησης ειρήνης. Πρόκειται για μια σφαιρική προσέγγιση την οποία και εσείς συζητάτε εκτενώς εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενισχυθεί περισσότερο ο διάλογος και η διαμεσολάβηση με διάφορες χώρες για να καταφέρουμε να έχουμε τελικά και αποτροπή των συγκρούσεων αλλά και ανοικοδόμηση αποκατάσταση των κοινωνιών και των κρατών που εξέρχονται από ένα πόλεμο, μια σύγκρουση. Έχει ήδη δημιουργηθεί και ένα γραφείο για, τον, για το μη αποκλεισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Καναδά. Προσπαθούμε μέσω του γραφείου αυτού να ελέγξουμε και τη δική μας την παρουσία σε διάφορες χώρες, εκεί πέρα που έχουμε αποστολές και Προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε ως Καναδάς πιο αποτελεσματικά στο πλευρό των εταίρων μας. Όπως σας είπα, ο Πρωθυπουργός μας ήταν εδώ πριν από 1,5 μήνα. Ήρθε όμως και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος συνάντησε την κυρία Μογκερίνη, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζήτηματα εξωτερικής πολιτικής και μου είπε ότι έχουν μια πάρα, ένα πολύ επικοδομητικό διάλογο, όχι μόνο επειδή έχουμε κοινέ προτεραιότητες, αλλά επειδή προσπαθούμε από κοινού να δούμε πώς μπορούμε να διαρθρώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνεργασία μας. Έχουμε από τη μία τη ΣΥΤΑ, και από την άλλη, όπω σα είπα, και αυτή τη συμφωνία στρατηγική εταιρική σχέση μα επιτρέπουν πλέον οι δύο αυτέ συμφωνίε να μπορέσουμε σε πολυμερέ και διμερές επίπεδο να συνεργαστούμε όλο και πιο αποτελεσματικά σε μεγαλύτερο βάθο. Από στρατιωτικής πλευρά, όπω σα είπα, έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία και νομίζω ότι τα πράγματα θα κινηθούν όλο και πιο αποτελεσματικά στο μέλλον. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκουμε εδώ πέρα σήμερα, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε μια πολύ θετική συνεργασία για ζητήματα ασφάλεια και προσβλέπω τώρα σε ερωτήσεις και παρατηρήσεις Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Βεβαίως όλοι έχουμε επίγνωση του πόσο μεγάλη είναι η σφορά του Καναδά στην ε, παγκόσμια ε, στρατηγική ασφάλειας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ αυτή την προχωρημένη ώρα και πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Καταρχήν θα ε, διατυπωθούν κάποιες ε, ερωτήσεις. Ο κύριος Γκάλερ, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρέσβη. Ε, πραγματικά είναι ένα προνόμιο και είναι μια καλή ευκαιρία να ακούμε τον πρέσβη μιας ε, φιλικής προς εμάς χώρας ε, και αν γνωρίζαμε ότι η χώρα σας ε, είναι βόρεια της Αμερικής, ε, εκεί που βρίσκεται γεωγραφικά, θα πιστεύαμε ότι είναι ευρωπαϊκή αυτή η παρουσίαση. Πραγματικά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές κοινέ αξίες, αρχές, συγκλίνουν η πολιτική αξιολόγηση και νομίζω ότι αυτές τις τόσο δύσκολες ε, μέρες ή μάλλον αυτές τις δύσκολες ε, εποχές ε, σε παγκόσμια κλίμακα είναι μεγάλη τύχη να έχουμε έναν τέτοιο εταίρο όπως εσείς και πιστεύω ότι αυτό είναι αμοιβαίο και ιδιαίτερως όταν πρόκειται για θέματα όπως αυτά τα οποία συζητούμε εδώ χαίρομαι που επαναλάβατε τη δέσμευσή σας σε σχέση με τη Ρωσία, την Ουκρανία και ε, άλλες ε, περιοχές όπου σοβούν ε, κρίσεις. Είναι σημαντική η καναδική παρουσία, για παράδειγμα στην Τινησία, εκεί όπου εσείς αρχικά είχατε κάποιες επιφυλάξεις uh, uh, και ε, στο να νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η συνεργασία με τον Καναδά ε, και αυτό είναι λιγότερο μια, μια ερώτηση ε, παρά είναι μια διαπίστωση σε σχέση με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση σε σχέση με τη Ρωσία και την Ουκρανία υπήρξαν ορισμένα ερωτηματικά, αλλά ορισμένες παρατηρήσεις του κυρίου Τραμπ όσον αφορά την αμερικανική δέσμευση εντός του ΝΑΤΟ. Ε, εγώ ελπίζω ότι το περιβάλλον, το πλαίσιο στη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ θα παραμείνει πιστό στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και στη γενική πολιτική γραμμή. Και, ε, αλλά στην κατεύθυνση αυτή όλοι οι άλλοι εταίροι μπορούν να, είναι, να εισφέρουν στη διατήρηση της παραδοσιακής αμερικανικής ε, προσέγγισης. Δεν γνωρίζουμε τι μας ε, περιμένει σε σχέση με τη νέα κυβέρνηση, αλλά θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε για την ε, καλή σας συνεργασία. Thank Σας ευχαριστούμε, κυρία ναι, όντω ήταν μια μεγάλη μέρα και περάσει η ώρα, αλλά είχαμε και αυτή την αποφράδα ημέρα, αλλά και σκοτεινή νύχτα που προηγήθηκε, όπως θα είπε πρόεδρο. Και για πετε μας, θα γίνει αυτός ο τυχό. Το ρωτήσανε. Ήταν υπόσχεση. Υποσχέθηκε τείχος στα σύνορα. Και λένε και για τον τείχο που θα χτίσει ο Καναδάς για να προστατευτεί από ό,τι προκύψει. Βέβαια συμφωνώ με όσα είπε ο Μάικλ. Βεβαίω και πολλοί θα προσπαθήσουν να κάνουν διόρθωση πορεία στον κύριο Τραμπ και στην πολιτική του. Το θέμα είναι πώ βλέπει κανεί τη σχέση με τι ε, Ηνωμένε Πολιτείε στο πλαίσιο που συζητούμε. Ανησυχεί ο Καναδά. Διάβαζα χθε το βράδυ. ότι τόσοι πολλοί υπέβαλαν αιτήσει για άδεια στον Καναδά ή για ε, παροχή, απονομή των πάντων ηθαγένεια. Τόσε πολλέ πολλέ ήταν αυτέ οι που έπεσε το σχετικό site τη κυβέρνηση. Σα είπε και ο Μάικλ, σα ρώτησε για τη Ρωσία. Εσεί τι συνέπειε, τι επιπτώσει βλέπετε να έχουν όλα αυτά για το ΝΑΤΟ. Οι δηλώσει Τραμπ ήταν πάρα πολύ επιβλαβείς για το ΝΑΤΟ. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα κατ' εσάς. Για τη Ρωσία τώρα συγκεκριμένα. Κάτι διάβασα το καλοκαίρι. Το συμπληροφορείο του Καναδά προειδοποίησε ότι θα έχει επιπτώσεις στην κυβερνοασφάλεια του Καναδά ο υβριδικός πόλεμος. Τέλος. Υπάρχει κάποιο τομέα όπου είναι εντυπωσιακή η δραστηριότητα του Καναδά, αξίζει του θαυμασμού μας η χώρα σας, το πώς τα καταφέρνετε καλά με το μεταναστευτικό. Αντίθετα από εμά. Με ασφάλεια και με νομιμότητα πλαισιώνεται αυτούς οι οποίοι είναι πρόσφυγες αυτοί οι οποίοι έτουν άσυλο, ούτως ώστε να μπουν στη χώρα νομίμως. Τους παίρνετε ουσιαστικά από την ανασφάλεια που βρίσκονται και τους φέρνετε στη χώρα. Ανοιχτή μεταναστευτική πολιτική, σοφή μεταναστευτική πολιτική. Οπότε υπάρχουν τώρα νομιμοί διάβλοι, ασφαλείς διάβλοι, Κάποιο να κάνει την αίτηση. Εμεί δεν τα κάνουμε όλα αυτά και με το που δεν τα κάνουμε, τι κάνουμε. Ενθαρρύνουμε, τροφοδοτούμε τα δίκτυα των διακινητών. Μου άμα πείτε πάνω σε αυτά δύο λόγια. Γιατί πρόκειται για μια πολύ θετική εμπειρία και για ένα παράδειγμα προ μίμηση που αποτελεί η χώρα σα. Ο κύριο Στάτινα. Σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ θετικό, κύριε Πρέσβη, που ήρθατε να μας μιλήσετε. Και μπράβο σας για την ευθύτα με την οποία ε, μας αντιμετωπίζετε. Καλά τα πει κυρία Γκόμες για την ανοιχτή σας πολιτική και προσέγγιση για το πώς καλοδέχεστε τους ε, πρόσφυγες από όπου αν προέρχονται. Έχω και πολλούς Τσέχους συμπατριώτες μου στη χώρα σας και κάποιος εξ αυτών ο κύριος Γέλινεκ, ο Σότο έγινε πρέσβης της χώρας μας και πρεσβευτής στον Καναδά. Έχουμε προσβήσει και από την Ουκρανία, ε, αναφέρθηκε ο αριθμός το 1,5 εκατομμυρίου και έχουμε και τους εσωτερικά εκτοπισμένους οι ο οποίοι βρίσκονται ακόμα στην ε, Ουκρανία. Φοβούμαι πως ότι καταστροφικό συμβεί στη χώρα πρόκειται να δημιουργήσει νέες ροές μεταναστών, νέες ροές προσφύγων προς την Ευρώπη ή και προς τον Καναδά. Επίσης μας μιλήσατε και για κυρώσεις. στον Καναδά κάποιο, ε, α πούμε, και ο Πρωθυπουργό. Έχει ασχοληθεί με το ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο ε, εις την συμφωνία του Μίνσκ, διότι θα πρέπει να βρεθεί μια εναλλακτική λύση από τη συμφωνία του Μίνσκ. Δεν μπορεί να θεωρείται ότι είναι σαν να μην υπάρχει η συμφωνία. Θα πρέπει κάτι να γίνει. Θα πρέπει να βρεθεί κάποιο εναλλακτικό σχέδιο. Δεν ξέρω, έχετε εσεί τέτοιο σχέδιο. Η πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα, και εγώ με τη σειρά μου να συμβάλλω στη συζήτηση γιατί θυμάμαι και πριν από 10 χρόνια τότε που Είχαμε διμερείς συνομιλίες με τον Καναδά. Ε, είχαμε κάποια κοινά προγράμματα τα οποία αφορούσαν την Ουκρανία. Οπότε και εμείς τότε μάθαμε πόσο άρτια ήταν η προσέγγιση πολιτική του Καναδά. Και ο Καναδάς και η Πολωνία Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να συσφιχθούν οι σχέσεις σας και η συνεργασία σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που ήταν σημαντικές αποφάσεις του Βίλνιους. Βέβαια, κρυμούν ακόμα αυτά τα προβλήματα και να δούμε τώρα πώς θα βοηθήσουμε την Ουκρανία, πώς θα σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες. Χρειάζονται κι άλλε μεταρρυθμίσεις. Μία μόνο ερώτηση εξοχότερα. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις σχετικά με την Αρκτική. Πώς βλέπετε τις ευρωπαϊκές προτάσεις όσον αφορά μια ε, γενική, ολοκληρωμένη στρατηγική. Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο. Αλλιώ απαντήσει ερωτήσει του αδέλφου. Ευχαριστώ, είναι εξαιρετικέ οι απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω για μία ακόμη φορά να είμαι σύντομο. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντως για τη συζήτηση αυτή που κάναμε και με μεγάλη χαρά θα επιστρέψω στην Επιτροπή σας για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Ιδίως αν δεν καταφέρω λόγω του περιορισμένου χρόνου να απαντήσω πλήρως σε ερωτήσεις σας. Κύριε Γκάλερ, καταρχά, χαίρομαι πάρα πολύ για τα όσα είπατε. Πολύ συχνά νιώθουμε κι εμεί οι Καναδοί Ευρωπαίοι. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το οποίο είπατε. Μα ακριβώ αυτό κάνει η ΣΥΤΑ, ακριβώ αυτό κάνει η στρατηγική εταιρική σχέση. Είναι, αν θέλετε, ό,τι πιο κοντινό μπορούμε να έχουμε στο να είμαστε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για την ίδια οικογένεια ουσιαστικά. Εγώ ερωτεύτηκα την Ευρώπη πριν από πολλά χρόνια ως μέρος και ως ιδέα και βέβαια ερωτεύτηκα και μία Ευρωπαία και την παντρεύτηκα και έχουμε δύο πολύ όμορφα τώρα παιδιά τα οποία είναι τόσο Καναδοί όσο και Ευρωπαίοι. Νομίζω ότι οι συμφωνίες αυτές θα επιφέρουν όχι μόνο μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και αξιωματούχων, αλλά θα φέρουν πιο κοντά και τους ίδιους τους πολίτες μας και θα δούμε περισσότερες τέτοιες ωραίες ιστορίες από τη δική μου. Αναφερθήκατε στην Τινησία καταπληκτικό παράδειγμα για την σχετική αυτή επιτυχία που θα πρέπει να δούμε στην ε, περιφέρεια αυτή. Χρειαζόμαστε την επιτυχία αυτή της ε, Τινησίας και χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργαζόμαστε Καναδάς και Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχείρηση αυτή της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν επικεφαλής. Βλέπουμε επίσης ε, στην ε, Βόρεια Αφρική αλλά και στη Μέση Ανατολή κάποιες περιπτώσεις όπου θέλουμε και εκεί να έχουμε επιτυχία, να σημειώσουμε επιτυχία. Η Τινησία πάντως είναι ένα πολύ θετικό παράδειγμα και πρέπει να επενδύσουμε στη χώρα αυτή περισσότερο. Αναφερθήκατε στο μέλλον, μάλλον στην θέση που κρατάμε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανία. Μπορεί να βασίζεστε σε μία συγκεκριμένη τοποθέτηση του Καναδά όσον αφορά το πρόβλημα αυτό. Θα έχουμε έναν διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία, αλλά θα συνεχίσουμε να έχουμε μια αυστηρή στάση απέναντι σε αυτή τη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ενωμένοι, Καναδά και Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη Ρωσία και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα συνεχή διάλογο μεταξύ ημών για το ζήτημα αυτό. Πολλά πράγματα μπορούμε να μάθουμε ένας από τον άλλον και μπορούμε από κοινού να αναλαμβάνουμε συνέχεια δράση. Και αν το κάνουμε αυτό θα είμαστε όλο και πιο δυνατοί. Άννα καταπληκτική καταπληκτική ερώτησή σας. Μακάρι να μπορούσα να απαντήσω σε όλε τι ερωτήσει σας. Πιστεύουμε πραγματικά στις ανοιχτέ κοινωνίες, στις ανοιχτέ αγορές. Είμαστε μια χώρα και το είπα αυτό και στα πλαίσια του ΣΥΤΑ. Έγινε μια πολύ μεγάλη ε, συζήτηση για μια συμφωνία εμπορική μεταξύ ΗΠΑ και Καναδάς δεκαετία του 80. Μπήκαμε τότε στην ιστορία του ΝΑΦΤΑ χωρίς να γνωρίζουμε εντελώ την επιφύλαση για τον Καναδά και σημειώσαμε και εκεί επιτυχία. Είμαστε μια χώρα που ανέκαθεν ήταν αναντιχτή στην μετανάστευση και γνωρίζουμε ακριβώς επειδή έχουμε μια εμπορική προσέγγιση, οικονομική προσέγγιση στα πράγματα, ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί προς τον έξω κόσμο. Και θεωρώ ότι μπορούμε να συμβάλλουμε από κοινού σε έναν πιο ειρηνικό κόσμο. Όσον αφορά τώρα τις Ηνωμένε Πολιτείες, τα σύνορα τα διαχειριζόμαστε πολύ καλά. Υπάρχει πλέον κοινή, ολοκληρωμένη διαχείριση των σύνορων μας με τις ΗΠΑ. Μπορούν οι πολίτες από τις δύο πλευρές να διέρχονται τα σύνορα αυτά χωρίς ε, ελέγχους. Προσπαθούμε πάντως στα πλαίσια του Καναδά να έχουμε ένα σύστημα κοινωνικό το οποίο να μοιάζει με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο ξέρουμε ότι συνάπτοντα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να έχουμε κοινά συστήματα όσον αφορά την ε, κοινωνία. Τώρα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, ακόμα και με το νέο καθεστώ του, παραμένουν ένα πάρα πολύ σημαντικό εταίρο. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Σίγουρα η σημερινή μέρα είναι πολύ δραματική, αλλά εμεί θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την επόμενη Αμερικανική κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργό μου προχώρησε σε δήλωση, όπω και πολλοί άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, και νομίζω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τι ευρείε αυτέ προοπτικέ που έχουμε με την Αμερική, το ότι έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινέ αξίε και στα πλαίσια του κοινού μα διαλόγου με σίγουρο θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινέ θέσει θα στεφθεί, πιστεύω, με επιτυχία και η μελλοντική μας συνεργασία με την Αμερική. Όσον αφορά τη Ρωσία, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, υβριδική πόλεμη, προφανώς τα φαινόμενα αυτά μας ενσυχούν πολύ. Γι' αυτό το λόγο χαρήκαμε πάρα πολύ για τη δήλωση που είδαμε στην Σύνοδο της Βαρσοβίας, η συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ σημαντική. Γίνανε δηλώσει και από πλευράς Καναδά την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν, για παράδειγμα, έχουμε στρατιωτικές δυνάμεις ε, που κάνουν ασκήσεις, καναδικές δηλαδή, στη Λετωνία, τότε περιμένουμε ότι όντω θα υπάρχει μια απόπειρα παραπλάνησης του κοινού και παραπληροφόρησης από την πλευρά της Ρωσίας. Βλέπουμε ότι πολλές φορές οι απειλές της Ρωσίας δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα των θεσμικών μας οργάνων και δοκιμάζουν ακόμα και την προσήλωσή μας σε κάποιες βασικές αξίες. Εγώ πιστεύω όμως ότι τα θεσμικά μας όργανα και οι αξίες μας είναι πολύ πιο ισχυρές από ό,τι τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Είναι ανθεκτικά λοιπόν. Μπορούμε λοιπόν μέσω των δοκιμασιών αυτών να βγούμε ακόμα πιο δυνατοί. Αυτό το είδαμε και στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική υπομονή, αν θέλετε, την οποία θεωρώ ότι διαθέτουμε. Είμαι αισιόδοξο αναγκαστικά από επαγγελματική πλευρά, αλλά είμαι και ειλικρινή σε αυτή την αισιοδοξία μου. Θα μπορούσα πολύ σύντομα να σα μιλήσω για το μεταναστευτικό μα σύστημα. Είμαστε εν γέννη μια ανοιχτή κοινωνία, όπω σα είπα ένα 1% του πληθυσμού μας κάθε χρόνο είναι βασικά πρόσφυγες οι οποίοι φτάνουν, 300.000 ανά έτος, μετανάστες και πρόσφυγες. Έχουμε μια πολύ αυστηρή επιτήρηση στο σύνορα μας και για αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους, ιατρικούς ελέγχους ή εγκληματολογικούς ελέγχους και όπως είπατε και εσείς τόσο ωραία έχουμε δημιουργήσει ασφαλείς νόμιμες οδούς για τη μετανάστευση. Οι περισσότεροι λοιπόν μετανάστες στον Καναδά μέσα σε τρία χρόνια γίνονται πλήρεις πολίτες του Καναδά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήδη υπάρχει ένας ομαλός δρόμος άφηξη και πρόσβασης των ανθρώπων αυτών στον Καναδά και στην αγορά εργασίας μας. Δεν είμαστε πολυπληθής χώρα, δημογραφικά δεν τα πηγαίνουμε τόσο καλά, υπάρχει υπογεννητικότητα, έχουμε και εμείς συγκεκριμένε ανάγκες. Επομένως, είμαστε μια ανοιχτή κοινωνία η οποία τιμά πραγματικά τα θετικά, τα ωφέλη της ε, πολυμορφίας, της διαφορετικότητας και φροντίζουμε κάθε φορά με τους μετανάστες να έρχονται μαζί τους και οι οικογένειές τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πραγματικά η ε, επιτυχής ένταξη στην κοινωνία μας έχει να κάνει και με το ότι οι μετανάστες ακολουθούνται από τις οικογένειές τους. Ξέρετε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή στον Καναδά για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου από τους πρόσφυγες και προσπαθούμε να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν πραγματικές ανάγκες, άνθρωποι που προέρχονται από καταβλισμούς όπως στο Λίβανο ή στην Ιορδανία, 40 με 50 χιλιάδες είναι ο συνολικός αριθμός των προσφύγων που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε υποδεχθεί στον Καναδά. Ξέρετε ότι οι πρόσφυγες είναι μια διαφορετική κατηγορία, συνήθως έχουν περάσει από τραυματικές ε, εμπειρίες, αλλά αν δούμε πραγματικά ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα που έχουμε όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα και όσον αφορά ακόμα και τα εισοδήματα, συνειδητοποιείται ότι αξίζει κανεί να κάνει μια επένδυση στου πρέσφυγε. Θα έλεγα ότι σε ορισμένε ευρωπαϊκέ χώρε γίνονται κάποια τέτοια πειράματα, μπορώ να τα αποκαλέσω έτσι. Κάθε χώρα όμω διαφέρει και δεν μπορούμε εμεί ω Καναδά να δώσουμε μαθήματα στου άλλου. Για παράδειγμα, ακόμα και ο ιδιωτικό τομέα ή πολλέ φορέ και οι οργανώσει εκπροσώπηση τη κοινωνία των πολιτών μπορούν να βοηθήσουν την ένταξη ορισμένων προσφύγων. Και νομίζω ότι αντίστοιχα παραδείγματα έχουμε και σε χώρε όπω η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αν δεν κάνω λάθο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχατε ανάλογε πρωτοβουλίε, όπω για παράδειγμα η πρωτοβουλία τη Μπλε Κάρτα. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τα απαραίτητα αυτά συστήματα που θα μα επιτρέψουν να προσελκύσουμε πρόσφυγες με συγκεκριμένες δεξιότητες. Εφόσον υπάρχουν όμως ήδη συγκεκριμένοι κανόνες σε μια χώρα, τότε η ένταξη των προσφύγων μπορεί να γίνει πιο γρήγορα και πιο ομαλά. Στην Σύνοδο Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε μία δήλωση. Σας παραπέμπω στη δήλωση αυτή όπου δεσμευτήκαμε να διερευνήσουμε έναν πιο ευρύ και σε βάθος διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη μετανάστευση. Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε ημένα από τους ΔΕ, από τη σωρευμένη εμπειρία μας και είμαι σίγουρος ότι μπορεί και ο Καναδάς να μάθει πάρα πολλά πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής ε, κρίσης. Να προχωρήσω τώρα παντώντας τον κύριο Τσέτνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναφερθήκατε στον κύριο Γέλνικ. Επέστρεψε στον Καναδά, αλλά πήγε πίσω και στην ε, Τσεχία, έτσι δεν είναι. Έχουμε ένα νέο πρέσβη τώρα, αλλά ξέρετε, άπαξ και είναι κανείς πρέσβης, παραμένει φόρου ζωής πρέσβης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αναφερθήκατε στην Ουκρανία, αναφερθήκατε στον Καναδά. Εγώ αναφερόμουν στον αριθμό των Καναδών που έχουν ουκρανική προέλευση. 1,3 εκατομμύρια είναι Καναδοί πολίτες οι οποίοι έχουν ε, καταγωγή από την Ουκρανία. Δεν πρόκειται δηλαδή για πρόσφυγες αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν και ένα εκατομμύριο Καναδοί οποίοι έχουν πολωνική καταγωγή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο του εθνικού μας ιστού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να κρατήσουμε μια κοινή ισχυρή στάση. Για παράδειγμα, στο Μίνσκ, η συμφωνία του Μίνσκ μάλλον, μπορεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή λύση, αλλά είναι η μόνη λύση που έχουμε αυτή τη στιγμή και θέλουμε να βοηθήσουμε τόσο την ομάδα της Νορμανδίας, όσο και τις προσπάθειες του ΑΣΕ. Αυτή τη στιγμή η συμφωνία του Μίνσκ ε, κατάφερε κατά κάποιο τρόπο να μειώσει το επίπεδο αιματοχυσίας, μόλον ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους στην Ουκρανία αλλά εφόσον είναι το μόνο πλαίσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, η συμφωνία του Μίνσκ, πρέπει να συνεργαστούμε στα πλαίσια τη συμφωνία αυτή. Και εμεί έχουμε πει ότι θα πρέπει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Καναδά να έχουν μία κοινή στάση, να μιλάνε με μία ενιαία φωνή όσον αφορά το ζήτημα τη Ουκρανία. Αυτό το έλεγα ανέκαθεν. Κυρία Πρόεδρε, απευθυνόμενο τώρα σε εσά και απαντώντα στις ερωτήσει σα. Θα ήθελα να πω ότι ξέρετε ότι ήμουν πρασβευτής στην Πολωνία και έχω ρωτευτεί και τη χώρα αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ για την πολύ θετική διμερή συνεργασία που έχουμε με την Πολωνία, η οποία άπτεται πάρα πολλών τομέων. Για παράδειγμα, στην Ουκρανία συνεργαστήκαμε πολύ στενά με Πολωνούς αξιωματούχους και πολωνικές στρατιωτικές δυνάμεις και έχουμε προσπαθήσει να προωθήσουμε μέσω της κοινή μας αυτής συνεργασίας τη δημοκρατία στη χώρα αυτή. Εκτιμώ ιδιαίτερα λοιπόν την συνεργασία που έχουμε με την Πολωνία όσον αφορά τις περιοχές του αρκτικού κύκλου. Ξέρουμε ότι με τις κλιματικές αλλαγές και με τις αυξανόμενες δραστηριότητες οικονομικές ε, στην Αρκτική, η περιοχή αυτή γίνεται μια περιοχή που είναι όλο και πιο προσβάσιμη τελικά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο καταβάλουμε και εμείς προσπάθειες προκειμένου να εμπλακούμε περισσότερο με τους εκεί ανθρώπους, με το γηγενή πληθυσμό, προκειμένου να γνωρίζουμε και ποια είναι η δική τους η άποψη όσον αφορά τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες. Και βέβαια συμβάλλουμε πάρα πολύ στο Αρκτικό Συμβούλιο και θα θέλαμε να επισημοποιηθεί το καθεστώς παρατηρητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αρκτικό Συμβούλιο. Το Αρκτικό Συμβούλιο αποτελεί ένα καταπληκτικό φόρουμ συζήτησης όλων των ζητημάτων που άπτονται της Αρκτική. Αναφερθήκατε επίσης στο ζήτημα της ασφάλειας στην Αρκτική. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν προβλήματα ή προκλήσεις ασφάλειας σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Πάντως εμείς θα παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις, όχι μόνο στη δική μας πλευρά του αρκτικού κύκλου, αλλά στον, στη γενικότερη περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουμε εκ των προτέρων ενδεχόμενες αναδυόμενες προκλήσεις. Θα έλεγα ότι η βασικότερη ανησυχία μας είναι να διασφαλίσουμε, πρώτον, ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνουμε έχουν ε, την έγκριση των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή εκεί και θα θέλαμε επίσης να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε ακόμα και με τη Ρωσία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αυτά θα έλεγα ότι είναι τα πιο ε, επίγοντα ζητήματα που μπορούμε ε, να εντοπίσουμε στην περιοχή αυτή. Προσβλέπουμε όμως σε περισσότερες συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίως στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αυτής προσέγγισης που θέλει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αρκτική. Ξέρω ότι ένα έγγραφο υποβλήθηκε επισήμως πριν από μερικές ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Είναι χαρά μας και προνόμιό μας να σας έχουμε εδώ ανάμεσά μας και ήταν πραγματικά μια αληθινή ευχαρίστηση να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε αυτή την τόσο φιλική ατμόσφαιρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ε, πρώτη μέρα της συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Ε, αύριο στις 9 ε, μας περιμένουν άλλα σημαντικά θέματα. Στις 9.30 σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξή μας. Ευχαριστώ πολύ.